After Μιας και έχει τόσο κόσμο μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα των έργων δημοσίων αστικών μεταφορών. Υπήρξε και μια σχετική έκθεση περιφερειακή έκθεση για 8 χώρες. Καταστροφική ήταν, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν τελικά χρήματα, τα οποία όμως ε, δαπανώνται με λάθος τρόπο, διότι υπάρχουν αεροδρόμια που υποδέχονται μία ή δύο πτήσεις τη μέρα. Προφανώς πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα και οπότε θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται και στις αστικές μεταφορές. Αν τα πράγματα είναι καλύτερα ή τα ίδια. Και χαίρομαι που είναι εδώ η κυρία Ιβανόβα από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα μας παρουσιάσει την συγκεκριμένη ειδική έκθεση. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σαν πρώην μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ υπό την ιδιότητά μου μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αναφερθώ στην έκθεση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της μεταφοράς στην Ευρώπη και παρουσιάζω τα συμπεράσματά μας στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Α, ελπίζω τα πορίσματά μας δεν θα φανούν τόσο άσχημα όπως ε, αναφέρατε για την προηγούμενη έκθεση. Να υπογραμμίσω γιατί επιλέξαμε το θέμα. Επελέγει το θέμα για έλεγχο από το συνέδριο υπό το φως του αυξανόμενου ε, Τη ευξανόμενης κέντρου του πληθυσμού σε αστικά κέντρα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία τα οποία μα δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συμφόρηση των μεταφορικών μέσων κοστίζει 80 δι ευρώ κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα τρία θανατηφόρα ατυχήματα συμβαίνουν σε αστικέ περιοχές. Η αστική κινητικότητα είναι υπεύθυνη για 23% των εκπομπών ε, διεξιδίου του άνθρακο στι οδικέ μεταφορέ. Η χορύπανση αυξάνεται σαν πρόβλημα στι ευρωπαϊκέ ε, πόλει. Και για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, στην περίοδο 2000-2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυσε 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ στις δημόσιες αστικές μεταφορές και προγράμματα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής. Οι κατασκευές, ο εξυγχρονισμός, οι επεκτάσεις υπογείου και διαφόρων μέσων ε, μεταφορών Συστήματα πληροφορικής υποστήριξης συμπεριλήφθησαν στις διάφορες χρηματοδοτηθήσει δράσεις. Γι' αυτό σχεδιάσαμε την έκθεση σαν έλεγχο επιδόσεων. Δεν εστιαστήκαμε επί των νομικών πτυχών ε, και τον του θεμητού χαρακτήρα των προγραμμάτων που συγχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογήσαμε την εφαρμογή τους και αποτελεσματικότητά του. Σε αυτό το πλαίσιο ασχοληθήκαμε με τα τρία βασικά ζητήματα τα έργα εφαρμόστηκαν όσοι είχαν σχεδιαστεί. Οι υπηρεσίες που παρεσχέθηκαν ε, κάλυπταν τις ανάγκες των χρηστών και χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα όσοι είχαν σχεδιαστεί και τα έργα. Λοιπόν, ε, διαλέξαμε πέντε κράτη-μέλη για να απαντήσουν σε ερωτήσεις Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία. Όλες μαζί χώρες καλύπτουν το 50% της συνολικής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης αστικές συγκοινωνίες την περίοδο 2000-2013. Εξετάσαμε 26 έργα, τα οποία όλα συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής κατά την λόγω περίοδο 2000-2013 και ίσως να είδατε στο παράρτημα 2 της εκθέσεως που διανύμαμε πριν την έναρξη της συνεδριάσεως αυτά τα στοιχεία. Ας εξετάσουμε εν συντομία τα πορίσματά μας εν γέννη. Τα περισσότερα έργα που ελέγχθησαν ή εφαρμόστηκαν και εκτελέστηκαν φυσικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Καθυστερήσεις επηρέασαν τέσσερα προγράμματα αστικών συγκοινωνιών. Υπήρξε ανάθεση ενός ελαφρού μετρό στην Πορτογαλία. Χρειάστηκε, ε, υλοποιήθηκε τρία χρόνια μετά την ημερομηνία που είχε προβλεφθεί. Η καθυστέρηση οφείλεται τις δυσκολίες να γίνουν η, να αγοραστεί η αναγκαία γη παρόλο που ήταν η διοκτησία των Δήμων. Διαπιστώσαμε επίσης ότι τρία έργα ε, ξεπέρασαν το προβλεπόμενο κόστος κατά σημαντικό πόσο. Επέκταση του μετρό στην Πολωνία ξεπέρασε κατά 22% την πρόβλεψη 47 εκατομμύρια που οφειλόταν σε σειρά δυσκολιών δυσμενείς συνθήκες ε, όσον αφορά το έδαφος. Όταν ολοκληρώθηκαν σχεδόν όλα τα έργα ε, εκάλυψαν τις ανάγκες των χρηστών. Στο έργο μας ε, τονίσαμε και τις καλές πρακτικές όταν υπήρχαν στην Πορτογαλία παραδείγματι. Βρήκαμε με τέτοια περίπτωση όπου η αμοιβή του φορέα που κινούσε του μετρό ανταποκρινόταν στις υπηρεσίες που παρήχε στους χρήστες καλή πρακτική. Αλλά το βασικό πόρισμα του έργου μας είναι τα δύο τρίτα των έργων ε, υποεχρησιμοποιούνται. Όπως θα βλέπετε και από το διάγραμμα 4 στη σελίδα 18, σε πολλές περιπτώσεις είχαμε μεγάλη διαφορά μεταξύ σχεδίου και της πραγματικής χρήσεως των διαφόρων έργων μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό σημαίνει υποεπίδοση όσον αφορά οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές στοιχές και ωφέλη όπως ε, μείωση της ρήπανσης και της συμφόρησης. Επιπλέον είδαμε ότι αυτά τα στοιχεία εν γέννη δεν ε, επαρακολουθούνται με τις εθνικές αρχές που ήταν επιφορτισμένες με τα έργα. Άλλο σημαντικό σημείο που θέλω να τονίσω ε, είναι οι συστάσεις μας Κατά την άποψή μα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διδραμάτισε σημαντικό ρόλο σχετικά με τα έργα. Τα περισσότερα είχαν ταξινομηθεί ε, ω σημαντικά έργα και ε, έπρεπε να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συστάσεις μας πρωταρχικά απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συγκεκριμένα συστήνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτεί ότι διαχειριστικά εργαλεία θα πρέπει να θεσπιστούν ούτως ώστε να υπάρχει παρακολούθηση της ποιότητας της υπηρεσίας και του επίπεδου ικανοποίησης των χρηστών από τη στιγμή που θα λειτουργούν πλέον τα έργα και τα... θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτεί ελάχιστο αριθμό δικτών αποτελεσμάτων που θα σχετίζονται με στόχους που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες χορηγήσεως χρημάτων και να υπάρχει η σωστή προσμέτρηση αυτών θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτεί να γίνεται μια εκτίμηση του αριθμού αναμενωμένων χρηστών ε, και να γίνεται καλύτερη ανάλυση αυτού του αριθμού και επιλογή του τρόπου μεταφοράς να στηρίζεται από ποσοτικοποιημένη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τρόπων ε, μεταφορών. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απαιτεί ότι τα προγράμματα αστικών μεταφορών να συμπεριλαμβάνονται σε μια γενική ε, πολιτική κινητικότητα. Συστήνουμε επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτεί από τις αρχές των κρατών μελών να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα όταν διαχειρίζονται ε, έργα αστικών μεταφορών, αστικών συγκοινωνιών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν εφαρμοστούν αυτά θα βελτιώσουμε και θα κάνουμε αποτελεσματικότερες ε, τις αστικές συγκοινωνίες στις ευρωπαϊκές πόλεις ε, ελπίζω ότι τα απορίσματά μας θα είναι χρήσιμα για το Ευρωκοινοβούλιο, κυρίως για τα μέλη της Επιτροπής αυτής, όπως ήταν χρήσιμα και για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών και προσβλέπω σε μια καρποφόρα ε, συζήτηση και ελπίζουμε πραγματικά να βοηθάμε όταν έρχεται η ώρα να πάρετε τις αποφάσεις σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Καλύτερα ακούγονται τα πράγματα από ότι με τα αεροδρομία. Βιν Βαντεκάμ έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μας χαρά να υποδεχόμαστε πρώην συναδέλφους Κάποιοι από εμάς Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι όταν έχουμε την ευκαιρία να πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο. Τρία σχόλια θέλω να κάνω. Πρώτον, νομίζω το κριτήριο της δημοκρατίας ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη το ελεγκτικό συνέδριο όταν ελέγχει τα θεσμικά όργανα. Επίσης μπορεί κανείς να δει την έκθεση αυτή με φιλικό ή όχι και τόσο φιλικό μάτι. Νομίζω ότι το ελεκτικό συνέδριο κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά είναι ε, πολύ σκληρή η έκθεση αυτή και όταν κάποιος ε, κατασκευάζει σύστημα μετρό ε, στην Πορτογαλία και τελικά δεν αξιοποιείται από τους επιβάτες, τότε συγγνώμη υπάρχει πρόβλημα. Η αντίδραση της Κομισιόν είναι σαφής, αλλά ελπίζουμε ότι θα εξαχθούν ε, και τα κατάλληλα συμπεράσματα ε, βάσει της συγκεκριμένης έκθεσης. Και το ερώτημα μου είναι προς το ελεγκτικό συνέδριο είναι μήπως, ε, μήπως είστε ευγενικοί σε αυτά που γράφετε ή τα πράγματα μήπως τελικά είναι πολύ χειρότερα από, από, από ό,τι καταγράφετε. Ευχαριστούμε Βιν Βαντεκάμ. Θέλω και εγώ να ακούσω την απάντηση, αλλά λίγη υπομονή χρειάζεται τώρα. Ο Ισμαήλ Έρτουγκ. Ευχαριστώ για την έκθεση αυτή. Σήμερα το πρωί ακούσαμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος τα πιθανά μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε και παρά το γεγονός ότι το θέμα ήταν ε, οι μεταφορές μεγάλων αποστάσεων ισχύουν παρόμοια πράγματα και στις αστικές μεταφορές. Και θεωρώ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει έλλειψη νομοθεσίας η οποία θα θεσπίζει ένα πλαίσιο για την συνύπαρξη των ε, κρατών Ξέρω ότι και στο Συμβούλιο έχουν εκφραστεί αντιστάσεις γιατί ορισμένες φορές το θέμα αυτό σχετίζεται και με ζητήματα επικουρικότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να σκεφτούμε αν τελικά θέλουμε να θεσπίσουμε νομοθεσία για τον τομέα αυτό. Γιατί σε τελική ανάλυση ισχύει ότι όσο πιο δίκαιη είναι η κατανομή του κόστους και αυτό αφορά και τις αστικές μεταφορές τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα. Εγώ δεν έχω ερωτήματα να θέσω αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι βέβαιος ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και ο νομοθέτης να καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ευχαριστώ, Λεπρόεδρος, για την Ευχαριστώ και εγώ για την έκθεση αυτή. Και εγώ χαίρομαι όταν ξαναβλέπω πρώην συναδέλφους, ιδιαίτερα όταν πλέον έρχονται με άλλη ε, ιδιότητα. Σε ό,τι αφορά την αστική κινητικότητα, νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα αυστηρούς νόμους, αλλά χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση ένα πλαίσιο για, την, ε, για τις αστικές μεταφορές και την ε, φιλικότητα προς, προς, προς το περιβάλλον. Υπάρχει, όπως είπε και ο Ισμαήλ Έρτουγκ, ε, η αρχή της επικουρικότητας, ενδεχομένως να υπάρχουν διάφορες, διαφορές όσον αφορά την, τις μεταφορικές υποδομές κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε όλοι ότι στις αστικές μετακινήσεις θα πρέπει και μπορούμε να γίνουμε πιο, ε, να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα, ε, γιατί τελικά Υπάρχει και το θέμα των ατυχημάτων. Στο Λονδίνο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εγώ έχω προσωπική εμπειρία ότι τα πράγματα λειτουργήσαν εξαιρετικά με, τους, ε, με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Οπότε το ερώτημά μου είναι, Ξέρετε ή θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες πόλεις ίσως θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρότυπα. Υπάρχουν κάποιες ε, πόλεις πρότυπα όπως ε, στην ε, Σουηδία από ό,τι ξέρω. Μπορείτε να μας δώσετε δηλαδή παραδείγματα αστικής μετα... αστικών μεταφορών που είναι και βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον και που εξυπηρετούν τους πολίτες τόσο στη δουλειά τους όσο και στον ελεύθερο χρόνο τους και όλα αυτά βεβαίως έχουν ωφέλη, και για το κλίμα και για την ποιότητα του αέρα στις πόλεις οπότε υπάρχουν κάποιοι φάροι ε, να το πω έτσι από τους οποίους θα μπορούσαμε να, ε, τους οποίους θα μπορούσαμε να μιμηθούμε επίσης νομίζω ότι θα χρειαστούν ενδεχομένως και κάποιες ε, διαφημιστικές εκστρατείες για συγκεκριμένους τρόπους μετακινήσεων. Δεν ξέρω αν γίνεται παντού, αλλά υπάρχουν ε, πόλεις στις οποίες, ε, για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν εναλλακτικά μέσα μετακινήσεων τι γίνεται με την ε, ηλεκτρική κινητικότητα, με τα ηλεκτρικά οχήματα. Το είπα και το πρωί ότι ε, βεβαίως σε αυτό το θέμα πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε και από πού προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια. Είπα το πρωί ότι στο Ανόβερο υπάρχει ένας σταθμός όπου μπορεί κανείς να φορτίσει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο και η ενέργεια προέρχεται από φωτοβολταϊκά που είναι εγκατεστημένα στο, στις ε, σκεπές αυτού του κέντρου και Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι αν υπάρχουν συνταγέ, αν υπάρχουν ωραία παραδείγματα, αν υπάρχουν θετικά παραδείγματα τα οποία ίσω θα μπορούσαμε να τα ε, κοινοποιήσουμε και σε άλλου για να τα μιμηθούν και άλλε πόλει. έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Euh, Σαν εισηγήτρια για την κινητικότητα την αστική στην Ευρώπη, θεωρώ ότι η αστική κινητικότητα είναι ή προκληστικός του πρωτεώνα γιατί, διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι 70% των πολιτών μας ζουν σε πόλεις και ότι οι πόλεις σήμερα δίνουν ε, τις δυνατότητες όσον αφορά την εργασία, την εκπαίδευση, πολιτιστικές δραστηριότητες και όσον αφορά την κινητικότητα. Και ότι υπάρχει αύξηση των περιβαλλοντικών πτυχών που λαμβάνονται υπόψη και αυξανόμενες ανησυχίες όταν μιλάμε για την αύξηση θερμοκρασίας, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ε, μέσω των πόλεων επηρεάζουμε το κλίμα, άρα είναι η πρόκληση του πρώτου αιώνα. Έχω κάποιες ερωτησούλες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξέρω αν κατά την απόψή σας υπάρχει αρκετή διαφάνεια όσον αφορά τα έργα αυτά. Δεύτερο ερώτημα ποια είναι η εξέλιξη της χρηματοδότησης των υποδομών είτε για τους ποδηλατόδρομους ή τη διαχείριση της κινητικότητας που θα έπρεπε να εφαρμοστούν. Θεωρώ ότι σήμερα η μεγάλη έλλειψη από τη συζήτηση είναι το θέμα της ήπιας κινητικότητας που είναι η συζήτηση επί της οποίας πρέπει να επιμείνουμε. Θα ήθελα να γνωρίζω επίσης Κατά την άποψή σας, ποια είναι τα εργαλεία για καλή διαχείριση αστική. Ποια είναι τα φημισμένα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουμε. Όλοι μιλούν για επικουρικότητα. Παραδείγματος χάρη, οι ακμές της μόλυνσης της πόλης σημαίνει ότι χρειάζεται σχεδιασμός της πόλης και οφείλεται στο σχεδιασμό. εάν οφείλεται στο ντίζελ και σε εκπομπέ σωματιδίων θα πρέπει να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αστική κινητικότητα σχετίζεται και με την αύξηση θερμοκρασία και με τον αντίκτυπο των νέων υποδομών. Τι είδου επενδύσει λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε, να δώσουμε. ποιε είναι οι αλλαγέ νοτροπίας που θα πρέπει να λάβουν χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα έθετα ένα ερώτημα ε, κάπως που ταιριάζει με αυτά που είπε ο κύριος Χέρτσογκ και δεν αφορά άμεσα την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Θα εκφράσω κάπως διαφορετική απόψη τον κύριο Χέρτσογκ. Ανακαλύπτοντας το θέμα, διερωτώ εάν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας η αστική συγκοινωνία συμπληρώνοντας αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο ε, κύριος Σαρτούκ σωστά αναφέρθηκε στην επικουρικότητα. Τι απομένει από την επικουρικότητα, τι μένει να αρμοδιότητα των κρατών μελών, για να το πω αλλιώ. Θεωρώ θεμητό η, Ευρωπα... Επιτροπή μας να ασχολείται με κάποια μεγάλα έργα υποδομών για τις μεταφορές που προορίζονται στη διασύνδεση χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεμητό να ασχοληθούμε παραδείγματι με συνδρομικές διασυνδέσεις τρένα υψηλή ταχύτητα ή εμπορευματικά τένα που συνδέουν Βόρεια και Νότια Ευρώπη. Όπως στην περιοχή του Λίγκυρα, όπως και σχέσεις με Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Ακόμα και αν επιφυλάσσομαι όσον αφορά τη σύραγγα που ε, συνδέει Λιόν και Τωρίνο παρόλο και αν που υπήρχαν παρεκκλήσεις που αναφέρατε κύριε Πρόεδρε, θέμητο να ασχοληθούμε με τα αεροδρόμια, κυρίως αν είναι διεθνή αεροδρόμια, από τα οποία διέρχονται αεροσκάφη που συνδέουν χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ευρωπαϊκή Ένωση με το εξωτερικό. Όμως, να ασχολούμεθα με τη χρηματοδότηση, στη χρηματοδότηση δύο χιλιόμετρων υπογείου στη Βαρκελόνη ε, σε, στη Βαλενσιένη, στην Χαύρη ή στη Φλωρεντία ή στην Κρακοβία νομίζω ότι αυτό δεν είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ρόλος των κοινοτήτων που είναι μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις, πλούσιες, που διαθέτουν τα μέσα και έχουν αναγκαία τεχνογνωσία και μπορούν να κρίνουν αν χρειάζεται να επεκτείνουν το δίκτυο του τραμ ή του μετρό. Και έχουν λύσεις εξαιρετικά διαφορετικές. Είναι ο ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν νομοί, τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ο ρόλος των κρατών μελών και όχι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτό αν θεωρούμε ότι η Ένωση θα πρέπει να διαχειρίζεται σε όλου του μετρο και εχουν λυσεις εξαιρετικα διαφορετικες ειναι ο ρολος τοπικης αυτοδικησης υπαρχουν νομοι τοπικη αυτοδικηση ειναι ο ρολος των κρατων μελων και οχι ο ρολος της ευρωπαικη ενωση εκτο θεωρουμε οτι η ενωση ζωή, τι μεταφορέ να μην μιλήσουμε για τον πολιτισμό, τη σεξουαλική ζωή. Να ελέγχει πλήρω τη ζωή 600 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. 500 ε, εκατομμυρίων Ευρωπαίων και αυτό το βρίσκω ότι είναι μια τρέλα πραγματική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, εγώ είμαι σκιώδη ε, η συγγήτρια και συμφωνώ με αυτά που είπε η Καρή Μαντέλη, ειδικότερα σε σχέση με τις προκλήσεις του 21ου αιώνα ε, το να δημιουργήσουμε δηλαδή πόλεις στις οποίες το μεγαλύτερο τμήμα ε, του πληθυσμού μας θα δει, να αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή, όπως επίσης να έχουμε μέσα μεταφοράς ασφαλή, ε, καθαρά, ώστε να μπορεί σε αυτό το περιβάλλον να ανθεί η οικονομία. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και ακόμη και μία μικρή στιγμή της, ε, μια μικρή απεικόνηση της καθημερινής κατάστασης δείχνει πόσο πολύ ε, δρόμο έχουμε μπροστά μας. Όσον αφορά τώρα το, την ανάλυση, νομίζω ότι καλώς ε, επικεντρωνόμαστε στη χρήση, όμως ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα θέμα με τα υπόλοιπα ωφέλη, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Καταλαβαίνω ε, αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με, με αυτά που είπε για τα μεγάλα προγράμματα υποδομής και ότι σε αυτά μερικές φορές δεν μπορούμε πάντοτε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι ειδικότερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους στόχους ασφάλειας, τη κοινωνική ενσωμάτωση, όλα αυτά τα πράγματα δεν εμφανίζονται σε αυτή την έκθεση και επίση αποδέχομαι το γεγονό ότι οι ελεγκτέ έχουν μια περιορισμένη εντολή, όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα καταφέρουμε καλά και να πετύχουμε μια ισορροπία. Και γιατί έχουμε διαλέξει αυτά τα πέντε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Αν δει κανεί τον πίνακα, τη σελίδα 7, ε, 6 και 7, το Ηνωμένο Βασίλειο λέει εδώ ότι έχει λάβει παραπάνω χρηματοδότηση από τα υπόλοιπα Καταλαβαίνω ότι απόψε ω ε, συνοχή μπορεί να είμαστε υποψήφοι για πιο πολύ χρηματοδότηση, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτό και για ποιο λόγο δεν, δεν αναφέρεται το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτά τα ε, πέντε κράτη-μέλη, τα 11 κράτη-μέλη ε, και έχω και σοβαρές ε, αμφιβολίες όσον αφορά τη ροή της χρηματοδότησης γιατί δεν γίνεται επαρκής δουλειά για να ε, συνοψιστούν όλα όπως πρέπει και όλοι οι εταίροι να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν τις ευκαιρίες αυτές για να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτό το σημαντικό θεματολόγιο. Η ανάλυση για την απορρόφηση είναι ένα θέμα το οποίο ε, το είχα θέσει και όταν ε, το ECA είχε κάνει την έκθεση πριν από μερικού μήνε ότι δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε πια στην απορρόφηση. Για ποιο λόγο να έχουμε αυτέ τι τεράστιε ροέ χρηματοδότηση αν δεν ε, χρησιμοποιούνται, δεν αξιοποιούνται οι απαραίτητε ευκαιρίε. Και νομίζω ότι η συγκεκριμένη έκθεση πρέπει να εδωθεί ω ως τμήμα του ευρύτερου προγράμματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σωσμπάχ. Ένα σύντομο ερώτημα για τις δημόσιες μεταφορές. Έχουμε κάνει πολλές φορές τις συζητήσεις για τις απευθείας αναθέσεις, για τους διαγωνισμούς και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αναλύσατε, αν εξετάσατε το συγκεκριμένο ερώτημα και αν ε, διαπιστώσατε ε, ότι, ε, ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων όσον αφορά ε, την συμμόρφωση, την αποτελεσματικότητα και τα Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και εν ώψη του τέταρτου πακέτου για τους σιδηροδρόμους. Εγώ είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων, δηλαδή οι δήμοι να έχουν βάσει της επικουρικότητας, της αρχής επικουρικότητας τη δυνατότητα να ε, επιλέγουν μόνα τους την, ε, ε, την ανάθεση έργων. Υπάρχουν όμως και κράτη-μέλη που ακολουθούν τη διαδικασία των διαγωνισμών και αν τέλος πάντων διαπιστώσατε εσείς να υπάρχουν διαφορές. Και εγώ έχω ένα ερώτημα. Κύριε Γκόλνης. Κύριε Γκόλνης. Αν κάποια πόλη, κάποιος δήμος δεν θέλει χρήματα ε, σε αυτές τις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρεμβαίνει, ούτε διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Αλλά αυτό που δεν γίνεται να δεχτούμε είναι να παίρνουν πόλεις λεφτά και μετά να μην θέλουν την παρέμβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το να, ασχοληθεί, το να ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αστικές μεταφορές είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν και οι στόχοι για το κλίμα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι στόχοι για το κλίμα είναι εξαιρετικοί, αλλά δεν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει στις αστικές μεταφορές, διότι οι αστικές μεταφορές ευθύνονται κατά 70% στις εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου. Χωρίς αλλαγή στις αστικές μεταφορές δεν πρόκειται να επιτύχουμε τους στόχους για το κλίμα. Όποιος λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτούς τους ε, στόχους, τότε πρέπει να παρέμβει και στις αστικές μεταφορές. Να σας πω τι έγινε στο Βερολίνο. Δέκα χρόνια μας ε, λέγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει χρήματα για αστικές μεταφορές, μόνο για αυτοκινητόδρομους. Εμείς θα θέλαμε, ε, λέγανε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο χαζή που δεν μας δίνει χρήματα ήταν ψέμα, κατάφορο. Και μάλιστα το είπε ο Υπουργό Οικονομικών του κρατηδίου και το τμήμα του, το, το επιτελείο του. Εγώ τον, ε, τον αποκάλυψα και το έβγαλα στη δημοσιότητα. Δεν είπαν συγγνώμη ποτέ. Γι' αυτόν τον λόγο, για τις αστικές μεταφορές, η Γερμανία απορρόφησε μέσα σε 10 χρόνια μόνο 62 εκατομμύρια ευρώ, παρά το γεγονός ότι είναι μεγάλη ε, χώρα. Αυτά να σας πω για, ως παράδειγμα για το πώς μπορεί να παρέμβει κανείς στις αστικές μεταφορές και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τότε θα έχει δικαίωμα, κάθε δικαίωμα να ε, παρεμβαίνει. Πορτογαλία, έχω ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα αυτή γιατί ε, γνώρισα και το τραμ γιατί οι δρόμοι είναι πάρα πολύ ε, στενοί και το τραμ, ε, ε, ο αστικός σιδηρόδρομος δηλαδή, ε, χρησιμοποιεί τους ίδιους δρόμους με τα αυτοκίνητα. Ε, χρηματοδοτούνται τέτοια έργα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί στην ε, Γερμανία δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση τέτοιων έργων γιατί υπάρχουν ε, ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών αυτοκινήτων. Για την ε, μη ικανοποίηση που ανέφερε ο κύριος Βαντεκάμ, μπορώ να πω ότι κατά 70-80% άκουσα Να ε, σας πω κάτι, το αεροδρόμιο του Βερολίνου κανείς δεν είναι μη ικανοποιημένος, δυσαρεστημένος, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Και αυτό κάτι λέει. Για την σιδηροδρομική σύνδεση Μπρέσλαου συνόρων υπήρξε συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον Γκέλ στο Βόρσα ε, επίσης ε, υπάρχουν ε, σιδηροδρομικές συνδέσεις. Ε, και αυτές τώρα καταργούνται τώρα αυτές οι συνδέσεις. Μήπως το ερώτημά μου είναι βρήκατε έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν αλλά τελικά δεν βρίσκονται σε λειτουργία γιατί κανείς δεν τα χρησιμοποιήσει. και επίσης θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα ποσοστά συγχρηματοδότησης, πόσο υψηλά είναι τα ποσοστά συγχρηματοδότησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με αυτό να περάσω στη σελίδα 18 και νομίζω ότι κάποιο λάθος έκανε εδώ ο Βιμ Βάντεκαμπ γιατί κάτω κάτω λέει 87% ε, λέει, αλλά αυτό δεν είναι το ποσοστό δυσαρέσκειας, είναι το ποσοστό κατά το οποίο επιτεύχθηκε ε, το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Είναι εξαιρετικός ο αριθμός αυτό, γιατί ειδικά αν ξέρει κανείς ε, αν έχει κάποιες γνώσεις για Τραμ γνωρίζει ότι χρειάζονται 2-3 χρόνια μέχρι να αξιοποιηθούν πλήρως και από τους επιβατητές. με 2 και 18% αντίστοιχα έργα στην Ισπανία βρίσκονται πολύ κάτω των προβλέψεων και αυτό που φαντάζομαι και υποψιάζομαι είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είχαμε τελικά να κάνουμε με συγκοινωνιακή πολιτική αλλά με εξυπηρέτηση των κατασκευαστικών λόμπι στο Βερολίνο, όταν έπεσε το τείχο, είχαμε τα ίδια προβλήματα με, άλλα, με, με, άλλες πόλεις. Γιατί είχαμε τραμ, 8 ε, γραμμές στο Ανατολικό Βερολίνο και ε, στο Δυτικό δεν υπήρχε. Αλλά για 5 χιλιόμετρα σε 30 χρόνια είχαν ε, δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για μετρό που θα μπορούσαν να είχαν κατασκευαστεί 120 χιλιόμετρα ε, τραμ και να σας πω θα ήθελα να μάθω πώς γίνεται αυτό και πώς εγκρίθηκε αυτό πώς είναι δυνατόν δηλαδή να, να εγκρίθηκε ένα τέτοιο έργο που απευθύνεται σε 2% τελικά των ε, πελατών των επιβατών δηλαδή στους οποίους απευθυνόταν Λοιπόν, επειδή μπλέκονται διάφορα και το τραπεζικό και το κατασκευαστικό λόμπι, θα ήθελα να τοποθετηθείτε και επ' αυτών. Και μια και δεν έχει ζητήσει κανεί άλλο το λόγο. Α, όχι, εντάξει, κατά εξαίρεση, νομίζω θέλει να. Κύριε Γκόλνη, θέλετε να απαντήσετε σε μένα, οπότε σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομη απάντηση. Καταρχά, να σα πω ότι τα τελευταία παραδείγματα που δώσατε πηγαίνουν προ τη δική μου κατεύθυνση. Είναι μια πάρα πολύ καλή απεικόνηση αυτή που κάνατε με αυτή την υπόθεση του μετρό στην Ιταλία δείχνει ότι οι κοινέ χρηματοδοτήσεις μερικές φορές δημιουργούν ανευθυνότητα. Καταλαβαίνω ότι είναι καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής θέρμανσης του πλανήτη αν οφείλεται βέβαια στην αύξηση του ποσοστού εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά η λογική αυτού του πράγματος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται τα, τις αστικές ζώνες και τις υποδομές τους και τις μεταφορές τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτρια. Δεν είμαστε καν σε μια ομοσπονδιακή κατάσταση. Πιστεύετε δηλαδή ότι η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες ασχολείται με τις αστικές μεταφορές, τη γεωργία, στην καλλιέργεια και στην Αλαμπάμα. Όχι, αυτό το αφήνει στα στις εν λόγω πολιτείες. Έτσι και εμείς προσπαθούμε ε, να κάνουμε το ίδιο. Εμείς δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να δημιουργήσουμε ένα ομοσπονδιακό κράτος λόγω του ότι υπάρχει κλιματική μεταβολή και θέρμανση του πλανήτη. Ωραία, ξανά έβαλα τον αυτό μου στον κατάλογο. Στον κατάλογο μιλητών ξανά έβαλα τον αυτό μου για να πω. Ε, η συγχρηματοδότηση είπατε ότι δεν είναι σωστή. Αλλά για, τον, ε, για το τραμ στην Πορτοβαλία εκεί που επιτέθηκαν 87% αυτή η συγχρηματοδότητα ήταν εξαιρετική γιατί η Πορτογαλία δεν θα μπορούσε να είχε επιτύχει ένα τέτοιο ποσοστό μόνη της. Να σας πω για την Αμερική. Ε, στη Βοστόνη ε, ο αυτοκινητόδρομος υπογειοποιήθηκε. Και αυτό έγινε γιατί το, η ομοσπονδιακή ε, κυβέρνηση ανέλαβε 80% του κόστους. Και αυτό λένε στη Βοστόνη οι άνθρωποι ότι οφείλεται στο όνομα του τότε κυβερνήτη της πολιτείας που τον έλεγαν Κέννεντι. Σας το λέω απλά σαν παράδειγμα για το πώς μπορεί η παρέμβαση από κεντρικούς φορείς να αλλάξει τα πράγματα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ε, προξένησα τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με την έκθεσή μου αυτή. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις του κυρίου Φαντενκάμπτ. Ε, κατά πόσο είμαστε φιλικοί ή μη φιλικοί, δεν νομίζω ότι προσπαθούμε να είμαστε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Προσπαθούμε να είμαστε εξισορροπημένοι και αντικειμενικοί. δεν προσπαθούμε να είμαστε καλοί, ό,τι βλέπουμε το λέμε, αν δεν δούμε τίποτε δεν λέμε τίποτα. Προσπαθούμε πάντως να δείξουμε τα θετικά παραδείγματα. Κάθε φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο είναι καλό νομίζω να ανταλλάσσουμε τις ε, καλές ε, πρακτικές και να τις ε, διαδίδουμε. Φυσικά θα επαφίεται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να μάθουν από τα λάθη που έγιναν και επίσης και από τις καλές πρακτικές. Όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις του Ισμαήλ Έρτογ, σε σχέση με το αν χρειαζόμαστε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, ε, αν πρέπει να υπάρξει νέα νομοθεσία δηλαδή, Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε δεδομένης της περιορισμένης ε, ε, εμβέλειας αυτής της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής θελήσαμε να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα, να μπορέσουμε να έχουμε ε, μετρήσιμους δείκτες για να δείξουμε και τα αποτελέσματα. Να συμπεριλάβουμε τα, τα προγράμματα αστικών υποδομών στην ε, πολιτική μεταφορών. Τώρα βέβαια αυτό είναι μια σύσταση για μας, ε, από πλευράς μας και για τα υπόλοιπα ερωτήματα νομίζω ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει κάποια από τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω εντός της ενός των αρμοδιοτήτων του ελεγκτικού συνεδρίου θα προσπαθήσω να απαντήσω στο δυνατόν περισσότερα ε, ερωτήματα. Κάποια άλλα πρέπει να τα απαντήσει η Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη συνάδελφο που έθεσε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της ε, βιωσιμότητας και βέβαια έχει να κάνει και με το προηγούμενο ερώτημα αυτό σε σχέση δηλαδή με την ε, ε, ανάγκη ύπαρξης λεπτομερέστερης νομοθεσίας και νέου νομοθετικού πλαισίου. Αυτό υποφύεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν εκείνοι θα αποφασίσουν να ακολουθήσουν την δική μας ε, σύσταση και να αναθεωρήσουν τις καλύτερες πρακτικές και να μπορέσουν να τις ε, ε, αποκρισταλώσουν σε μια νέα πρόταση για τις διαφημιστικές εκστρατείες ή οποιασδήποτε άλλες ε, ιδέες ή εμπειρίες υπάρχουν στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιηθούν αυτές και να διαδοθούν. Όσον αφορά την κυρία Ντελή, Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αυτή είναι η πρόκληση του αιώνα και η περιβαλλοντική διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε αρκετή διαφάνεια για τα προϊόντα, για τα προγράμματα αυτά. Ναι, παρακαλώ να θυμάστε ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των κρατών μελών, είναι πέντε. Για τον αριθμό των προγραμμάτων δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα πρόσβαση σε πληροφορίες δεδομένα. Βεβαίως αυτό δεν είναι οικονομικός έλεγχος, ο ετήσιος έλεγχος μας, η ετήσια μας έκθεση που αναλύει την ε, ορθότητα των συναλλαγών και της εφαρμογής και λοιπά είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ ασχολούμαστε μόνο με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των προγραμμάτων Τώρα όσον αφορά το επίπεδο ηχορύπανσης και τι πρόγραμμα έχουμε, πράγματι και εμείς θέλουμε να ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ποια ε, είναι η άποψή της για τη νέα νομοθετική περίοδο. Εμείς έχουμε υποβάλει τις συστάσεις μας και επ' αυτού και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και για τις βέλτιστες πρακτικές. Τώρα, για τα προγράμματα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη. Ε, αυτό ετέθη πολλές φορές, οπότε θα επανέλθω σε αυτό το θέμα και μάλιστα φτάνω έτσι στο σχόλιο του κυρίου Γκόλνης για την αρχή της επικουρικότητας και το ρόλου των κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που μπορούμε να πούμε βάση της περιορισμένης, του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής αυτής της έκθεσης ε, για την προγραμματική περίοδο όλα τα προγράμματα είχαν ταξινομηθεί ως μεγάλα προγράμματα. Πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ ήταν το κόστος τους. Αυτά που ήταν κάτω από τα 50 ε, εκατομμύρια εγκρίνονταν από, τη, από τα κράτη-μέλη. Στο παράδειγμα 2 της τελευταίας στήλης του πίνακα δείχνει, βλέπουμε ποια ε, προϊόντα ε, ελέγξαμε και ποια ενεκρίθησαν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα πώς θα είναι τα πράγματα για τη νέα προγραμματική περίοδο και εμείς έχουμε την απορία να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πάντως ε, οι αλλαγές προβλέπουν τα μεγάλα προγράμματα ε, θα δίνουν δύο επιλογές στα κράτη-μέλη. Ή θα υποβάλουν τα προγράμματα ως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα ε, δίνονται σε εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Στη δεύτερη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει έναν πιο περιορισμένο ρόλο, απλώς δηλαδή σιωπηλά θα εγκρίνει τα προγράμματα, εφόσον το καθήκον θα το έχουν οι εμπειρογνώμονε, αλλά αν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει περισσότερα γι' αυτό, ευχαρίστω. Εμεί αυτά γνωρίζουμε για την ώρα. Δεν ξέρουμε ποιε θα είναι οι αλλαγέ και θα, μας, θα, περιμένουμε κι εμεί να δούμε πώ θα γίνει στην πράξη η εφαρμογή. Κυρία Άνες, Άντερσον. Μιλήσατε κι εσείς για το θέμα της μεγάλης αυτής πρόκλησης. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη ε, για και για τα πορίσματά μας. Θα ήθελα να τονίσω σε σχέση με αυτά που είπατε ότι είναι περιορισμένη αυτή η έκθεση. Κοιτάξαμε τα επίπεδα ε, χρήσης, αξιοποίησης ε, ε, και τη μείωση της συγχωρήπανσης και τη μείωση και τον, την κοινωνική ενσωμάτωση που προκύπτουν έμεσα από τα πορίσματά μας. Για ποιο λόγο επιλέξαμε τα πέντε αυτά κρατημέλη. Εξήγησα ότι 50% των ποσών που διατέθηκαν ε, αφορούσαν τα 5-7 κρατημέλη. Ναι, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει και αυτό ένα μεγάλο ποσό, αλλά δεν είναι το υψηλότερο ποσό. Όταν διαλέγουμε τα κράτη-μέλη προσπαθούμε να δούμε και θέματα όπως η γεωγραφική κατανομή. Τα κράτη-μέλη δηλαδή που απορροφούν περισσότερα, γι' αυτό ακριβώς επιλέξαμε τα 5 αυτά να δουμε και θεματα οπως η γεωγραφικη κατανομη τα κρατη μελη δηλαδη που απορροφουν περισσοτερα γι αυτο ακριβως επιλεξαμε τα πεντε αυτα κρατη μελη και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μικρότερος δικαιούχος ε, εμπροκειμένου σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη. Ε, το θέμα τώρα που θέσατε για την απορρόφηση και τη χρήση της χρηματοδότησης αυτής, αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό απλώς να χρησιμοποιούμε, να ξοδεύουμε λεφτά απλώς και μόνο για να ξοδεύουμε λεφτά. Είναι σημαντικό να ξέρουμε και γιατί τα ξοδεύουμε ε, και τι προκύπτει από αυτή τη χρηματοδότηση, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο βασικός στόχος της δικής μας έκθεσης επιδόσεων, να δείξουμε τα αποτελέσματα και πώς άλλαξε η ζωή των Ευρωπαίων συμπολιτών μας ε, αν άλλαξε προς το καλύτερο πόσο επιτυχείς ήμασταν ε, ως προς αυτή την πτυχή της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Ο κύριος Μπαχ μας μίλησε για τις δημόσιες προμήθειες. Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν είναι τμήμα του συγκεκριμένου ελέγχου, αλλά Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή μία μελέτη που θα αφορά συγκεκριμένα το θέμα των δημοσίων προμηθειών. Θα δημοσιευθεί σύντομα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τμήμα της έκθεσης που παρουσίασα σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, Νομίζω ότι απάντησα την ερώτηση του ποιο εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μεγάλα προγράμματα για αυτή την προγραμματική περίοδο και τις αλλαγές που θα γίνουν από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Όσον αφορά το ήπιο μετρό, το κατά πόσο θα το κάναμε αυτό στη Γερμανία, ρωτήστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν αποφασίζει το ελεγκτικό συνέδριο γι' αυτό. Όσον αφορά τώρα το ποσοστό συγχρηματοδότησης, μπορούμε νομίζω να βρούμε την απάντηση στις σελίδες 26-27, όπου αναφέρεται ο κατάλογος όλων των ε, προγραμμάτων που ελέγχθησαν. Ε, βλέπετε ποιος έκανε την έγκριση, ποιο ήταν το κόστος, ποιο ήταν το συνολικό κόστος και από πότε ήταν ε, ε, επιχειρησιακό. Δεν μπορώ να πω τίποτε παραπάνω από αυτά που, έχω γράψει, που έχουν γραφτεί σε αυτή την έκθεση και που είναι ε, ε, δημόσια. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Ναι, αλλά δεν μου απαντήσατε το 87% των πελατών. Το 87% είναι το επίπεδο πρόβλεψης. Συγγνώμη, ναι, αυτό δεν το, δεν το απάντησα όντω. Για την Πορτογαλία, 87% των χρηστών ήταν ικανοποιημένοι. Να το επαναλάβω. Ευχαριστώ Βίμ βέβαια για τον καφέ, αλλά θέλω να το ξανατονίσω. 87% ήταν το υψηλότερο ποσοστό από αυτά που ε, σύμφωνα με, το, με τις προβλέψεις. 87% επετεύχθη λοιπόν και στο, στα μετρό. Στην Ιταλία για παράδειγμα επετεύχθη, μόνο, μόνο το 2% των, ε, των όσων προβλέπονταν δηλαδή των, με βάση τις προβλέψεις. Επίσης ξέχασα να αναφέρω τα καλά παραδείγματα, τα θετικά παραδείγματα που προσπαθώ πάντοτε να το κάνω υπήρξαν και σχετικές ερωτήσεις και έχουμε στον πίνακα 5 στη σελίδα 17 δύο έργα για τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας ε, δεδομένα και στοιχεία, έργα τα οποία επέτυχαν τους ε, στόχους για τους οποίους υλοποιήθηκαν. Είναι λοιπόν μια βέλτιστη πρακτική την οποία μπορεί κανείς να την κοινοποιήσει. Να κάνω μια συνόψη, ε, να συνοψίσω λίγο την συζήτηση. Ε, προς την Κομισιόν, σας παρακαλώ. Να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Το να κατασκευάζεται γραμμή μετρό που καταλήγει να ικανοποιεί μόνο το 2% των όσων, ε, ε, των όσων σκόπευε να ικανοποιήσει ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ότι μπορούν να χρτιστούν με τα χρήματα αυτά 57 ε, χιλιόμετρα ε, γραμμών τραμ, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν κάποιος αιτείται την κατασκευή τέτοιων έργων. Παρακαλώ κάθε φορά ενδελεχής ε, έλεγχος και να το έχετε υπόψη σας αυτό. Ένα λεπτό, αν επιτρέπετε, εφόσον ενδιαφέρεστε για το έργο μας, δάτω τι ευκαιρίες να ανακοινώσω ότι έχουμε και άλλη μελέτη που εμπίπτει στο πεδίο που σας ενδιαφέρει η έκθεση για διαδρομές εσωτερικής ναυσιπλοείας, αποτελεσματικότητα αυτών και άπτεται των ερωτημάτων του κυρίου Γκόλνιτς και των θεμάτων που έθιξε περί συντονισμού, περί γενικού στρατηγικού προβληματισμού για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Αν ενδιαφέρεστε με τα χαρά σας παρουσιάσω και αυτή την έκθεση σύντομα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Can you please... Βάντερ Κάμπ, Μπορείτε να μας πείτε πότε θα είναι έτοιμη αυτή η έκθεση όσον αφορά τις οδούς εσωτερικής ναυσιπλοείας. Από ό,τι κατάλαβα είναι έτοιμος. Σε κάνα δύο εβδομάδες θα δημοσιευθεί. Μετά από αυτό, από σας εξαρτάται. Αν ολοκληρωθεί, γνωστοποιήστε το μας. Να είναι πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Θα το κάνουμε, έτσι θα κάνουμε μάλιστα. nicht dabei ist, kann es eigentlich nur positiv sein τελικά έτσι έχουμε θετικές εξελίξεις. Λοιπόν, και τώρα νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε κάποιο χρόνο πριν το επόμενο σημείο. Α, είναι όλοι εδώ. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. So, dann können wir zum nächsten Ωραία, περνάμε στο επόμενο θέμα της ημέρας διάταξης. Παρουσίαση της έκθεσης Κριστόφερ Μπόντεβιξ έχει σχετικά με τα νέα χρηματοδοτικά συστήματα για έργα υποδομής στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών και στο πλαίσιο του ε, ε, Υπουργείου του, του Άτυπου Συμβουλίου η Ιταλική ε, Προεδρία ε, σε συνεργασία με τους ε, δύο Ευρωπαίους ε, συντονιστές, τον κύριο Μπόντεβι και Σέικη, κάλεσε να υποβάλει έκθεση για τα νέα χρηματοδοτικά συστάματα. Και αυτή η έκθεση παρουσιάστηκε στους Υπουργούς Μεταφορών. Τα απορίσματα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα όσον αφορά το, το εν και του, της ανάπτυξης του Ταμείου Στατηγικών Επενδύσεων του γνωστού ως σχεδίου Juncker. Γι' αυτό χαιρόμαστε που είναι εδώ οι τρεις κύριοι αυτοί. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοφόρου. Οπότε ε, δίνω πρώτα απ' όλα το λόγο στον κύριο Κριστόφερσεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. I'm here accompanied Είμαι εδώ συνοδευόμενος, όπως είπε ο Πρόεδρος, από τον κύριο Μπόντεβι από εδώ, από δεξιά μου λέει ο μιλητής, και δίπλα του έχουμε τον καθηγητή Κάλος έτσι από την Ιταλία. Συνεργαζόμαστε. Επεξεργαζόμαστε την τελική έκθεση που μας ζήτησαν οι Υπουργοί Μεταφορών στο Μιλάνο. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε έτοιμη την έκθεση πριν το τέλος της Λετωνικής Προεδρίας. Άρα αρχές Ιουνίου και μπορεί να μπει και στη γενικότερη συζήτηση για το πακέτο Juncker. Είναι ένα κομμάτι της δουλειάς που ζητήθηκε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μέχρι τώρα παρουσιάσαμε μια διάμεση έκθεση, όπως είπε σωστά ο Πρόεδρος. Ήταν αρκετά ευπρόσδεκτη από τους υπουργούς Μεταφορών στις 3 Δεκεμβρίου και χαίρομαι που είμαι εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών του Κοινοβουλίου και θα αναφερθώ εκτενέστερα στο γιατί είμαι ικανοποιημένος γι' αυτό. Το έργο της έκθεσης, όπως είπε ο Πρόεδρος, ακολουθεί το άτυπο Συμβούλιο Μεταφορών της 16-17 Σεπτεμβρίου του 2014 που έγινε στο Μιλάνο. Εκεί μαζί της Ιταλική Προεδρία στο Συμβούλιο και ο Επίτροπος ο κ. Κάλλας μας ζήτησε να ετοιμάσουμε μια έκθεση εντοπίζοντας προγράμματα, διαδρόμους καινοτόμα προσέγγιση στα πλαίσια των προσπαθειών για ανάπτυξη θέσης και επενδύσεις και το σχετικό πακέτο που είχε προτείνει ο πρόεδρος Γιούγκερ. Κάτι που έγινε δεκτό θετικά από το Κοινοβούλιο, όπως το εκλαμβάνω και είναι κάτι που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών. Στέρεη βάση δηλαδή. Να πω μερικά λόγια όσον αφορά τη φύση της έκθεσης. Δεν είναι έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε καλή κατανομή καθηκόντων μεταξύ μας, αλλά είναι μια έκθεση και των τριών και πρέπει να ακούσετε τις απόψεις μας σαν προσωπικές απόψεις. Συμβάλλει στη συζήτηση αυτή η έκθεση όσον αφορά το επενδυτικό πακέτο. Και ο δόκτωρ Μπότεβιτ και ο καθηγητής Σεκί αργότερα θα προβούν σαν ανάλογες παρουσιάσεις που αφορούν τμήματα της έκθεσής μας. Βασικός στόχος είναι να εντοπίσουμε προγράμματα όσον αφορά τους διευρωπαϊκούς διαδρόμους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια καινοτόμων χρηματοπιστωτικών πλαισίων. Είναι αναγκαίο, το γνωρίζουμε, ότι τα κάτι μέλη δεν έχουν μεγάλα πλεονάσματα ούτε διαθέσιμους πόρους για τέτοιου είδους επενδύσεις. Αντιθέτως μάλιστα, τα περισσοτερα κάτι κράτη-μέλη βρίσκονται σε μια κατάσταση στην οποία πρέπει να ψάξουν να βρουν άλλες πηγές χρηματοδότησης. Μία λύση θα ήταν να δούμε κατά πόσο μπορεί να ε, εμπλακούν οι ιδιωτικοί επενδυτές, όχι να διονοδοτήσουν, να γίνουν συνεπενδυτές, να αναλάβουν κάποιο κίνδυνο, να μοιραστούν τον κίνδυνο με δημόσιους φορείς και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους δανειοδότες. πέραν αυτού. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στην ομάδα μας θεωρήσαμε ότι υπάρχει ανάγκη να εντοπίσουμε τις αναγκαίες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ούτω ώστε να εξασφαλίζουμε αντιστοιχεία μεταξύ προγραμμάτων που απαιτούν επενδύσεις και των επενδυτών που προσπαθούν να βρουν επενδυτικές ευκαιρίες. Το λέω αυτό διότι κάπου ακούστηκε να λέγεται ότι αυτοί οι άνθρωποι στη Γενική Διεύθυνση για τι μετακινήσεις δεν ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα Juncker, το σχέδιο Juncker. Αντιθέτως, ελπίζουμε να είναι πολύ επιτυχές αυτό το πακέτο. Δημιουργήθηκε μεγάλη αισιοδοξία από την παρουσίαση του σχεδίου. Όμως βλέπουμε κάποια εμπόδια για την υλοποίηση του σχεδίου Πρέπει να γίνουν πρώτα κάποιες εθνοτικέ αλλαγές. Αυτό είναι έργο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των θεσμικών τη οργάνων. Είναι έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου των Υπουργών, επεξεργαζόμενοι την πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να επιτύχουμε και γι' αυτό με λίγα λόγια θα προσπαθήσω να σκιαγραβήσω το αποτέλεσμα της, ε, που αναφέρεται στην ενδιάμεσή μας έκθεση ο θετικός αντίκτυπος των επενδύσεων για τις υποδομές, για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα θα αναφερθούν από τον κύριο Μπόντεβιτς. Εγώ δεν θα πω πολλά, όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά για οικονομική ανάπτυξη, τα δίκτυα τα μεταφορικά, για δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ενιαία στέρεη επενδυτική στατηγική, διότι είδαμε δυστυχώς μεγάλη μείωση των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 5-6 χρόνια. Αυτές οι επενδύσεις δεν, σχε... σχετίζονται μόνο με την κατασκευή υποδομών που λείπουν, αλλά είναι σημαντικό οι επενδύσεις να χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των υφισταμένων δικτύων. Διότι έχουμε δαπανίσει 30-40 χρόνια για να κατασκευάσουμε αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια κλπ. στην Ευρώπη. Και αν δείτε ποια είναι η ποιότητα των δικτύων, θα διαπιστώσετε ότι χρειάζονται συντήρηση και αναβάθμιση και εξυγχρονισμό. Δεν χρειάζεται εδώ να σας μιλήσω για τους γαλλικούς αυτοκινητοδρόμους, τους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους. Όμως υπάρχει πραγματικά ανάγκη συντήρησης των δικτύων και χρειάζεται να έχουμε και κατάλληλα συστήματα μεταφορών για να χρησιμοποιούμε καλύτερα τις υποδομές και να χρησιμοποιήσουμε και τις αναγκαίες τεχνολογίες για καθαρές μεταφορές στα οχήματα και στις υποδομές η προσωρινή αυτή έκθεση παρέχει παραδείγματα έργων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τα σχήματα αυτά και τα σχέδια τα χρηματοπιστωτικά. Εστιαστήκαμε επί της ανάγκης να δημιουργήσουμε σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις. Να μιλήσουμε σε εκείνους που επενδύουν στα προγράμματα και σε εκείνους που προωθούν τα διάφορα έργα. Εντοπίσαμε διάφορα εμπόδια που εμποδίζουν τους ιδιωτικούς επενδυτές και έτσι δεν θέλουν να ψάξουν να βρουν επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα αυτό. Και μπορούμε να περιγράψουμε στην έκθεση τι μπορούμε να κάνουμε να γίνει πιο ελκυστικό ο τομέας για ιδιωτικούς επενδυτές. Όμως, είμαι αισιόδοξο ταιριάζουν οι οικονομικές ανάγκες των μεταφορικών υποδομών και των σχετικών έργων με το είδος των επενδύσεων που εξετάζουν οι θεσμικοί επενδυτές, όπως ταξιδιωτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείε. Και επίσης ο χρονικός ορίζοντας για τους χρηματοπιστωτικούς φορείς ταιριάζει με το χρονικό ορίζοντα για τη χρηματοδότηση και αποπληρωμή πολλών επενδύσεων που χορηγούνται για τις υποδομές όμως το ποσοστό ιδιωτικών επενδύσεων υποδομές περιορίζεται λόγω φραγμών. Να αναφέρω κάποια από τα εμπόδια. Υπάρχει έλλειψη σαφούς τρόπου δρομολογήσεως των προγραμμάτων. Αυτά που έχουμε δρομολογήσει δεν αρκούν. Υπάρχει έλλειψη σαφούς και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου σε κάποιους τομείς. Παραδείγματο χάρη όσον αφορά τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Τι αποτελεί κρατική ενίσχυση. Σε ποιο βαθμό είναι δυνατό να χορηγηθεί κρατική ενίσχυση. Τι γίνεται με διασταυρούμενη επιδότηση όταν επενδύει σε συνδυασμό σιδηροδρόμου και αυτοκινητοδρόμου και χρησιμοποιεί ένα τμήμα των εσόδων από το αυτοκινητόδρομο για να χρηματοδοτήσει τον σιδηρόδρομο. Σε ποιο βαθμό αυτό είναι δυνατόν. Τι γίνεται όσον αφορά διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει. Δίνει στο Κούκενχάβεν και όχι στο Βίλχεμσχάβεν ενίσχυση. Ή σε κάποιο λιμάνι και όχι στη Μασαλία Χρειάζονται διευκρινήσεις όσον αφορά τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Μετά, η συμπερίληψη των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και πώς συμπεριλαμβάνονται στο κρατικό χρέος. Πώς θα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη το Eurostat για να μην υπάρχει σύγκρουση με τα κριτήρια του Μάστριχτ ή με το πακέτο ανάπτυξης σταθερότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με το Βροστάτη αυτό. Υπάρχουν και έλλειψη κινήτρων για κάποιους θεσμικούς επενδυτές να επενδύσουν σε υποδομές. Διότι θεωρούνται σαν επικίνδυνες υποδομές όσον αφορά τη φερεγγιότητα. Και είναι και το θέμα της συντήρηση των υποδομών που δημιουργεί κινδύνου. Και θέλουμε να εξετάσουμε κάποιου τομεί. Δεν λέω θα υπάρξουν προβλήματα. Θα ελέγξουμε κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Έχουμε του κανόνες περί δημοσίων προμηθειών, αν λειτουργούν σωστά, αν επικρατεί επαρκή διαφάνεια, τα κριτήρια κατανομής είναι σωστά, οι διαδικασίες επιλογής προσφορών είναι αρκετά καλές. Έχουμε την αξιολόγηση επιπτώσεων για το περιβάλλον, τη σχετική διαδικασία λειτουργεί αρκετά καλά. Δεν έχω συγκεκριμένες παρατηρήσεις επ' αυτού. Ξέρουμε ότι χρειάζεται πολύς χρόνος να γίνει αξιολόγηση επιπτώσεων για το περιβάλλον. Καμιά φορά χρειάζεται χρόνος και για μικρά έργα, καμιά φορά είναι δαπανηρό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Έχουμε διαδικασίες για την αδειοδότηση κατασκευών. Είναι καλές. Μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα ενία θηρίδας. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να βελτιώσουμε την οριμότητα των έργων. Είναι το θέμα της δημιουργίας νομικών πλαισίων για τις συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα, πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι ιδιώτες επενδυτές και πώς μπορούν να επηρεάσουν τα έργα αν οι ιδιώτες αναλαμβάνουν κινδύνους. Πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν. Οι δύο συνάδελφοι θα αναφερθούν εκτενέστερα σε όλα αυτά. Είπα στην αρχή ότι χάρηκα που ήρθα εδώ και είμαστε όλοι μας χαρούμενοι που ήρθαμε εδώ. Διότι εμείς οι τρεις δεν έχουμε αρμοδιότητα να διαμεσολαβούμε μεταξύ των υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να διαμεσολαβήσουμε μεταξύ των κρατών μελών, μπορούμε να εντοπίσουμε προβλήματα, μπορούμε να εντοπίσουμε ευκαιρίες, αλλά χρειαζόμαστε πολιτική απόφαση ούτω ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει. Γι' αυτό είναι σημαντικότατο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι έτοιμο να επομιστεί τις ευθύνε του και να πει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τώρα πράγματα, υπάρχουν πράγματα πρέπει να γίνουν διότι δημιουργήθηκε μεγάλη αισιοδοξία από το πακέτο Γιούνκερ. Λοιπόν, αν αποτύχει, ίσως να έχουμε απρόβλεπτες πολιτικές συνέπειες. Σχετικά με αυτό, εμείς οι τρεις θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικότατο όχημα και ελπίζουμε ότι αργότερα θα μπορέσουμε να επανέλθουμε και να παρουσιάσουμε τα τελικά μας πορίσματα και μετά να δούμε πόσο επιτυχής θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, πώς θα εφαρμόσουν τις αναγκαίες προσαρμογές. Και εδώ να δώσω το λόγο στον δόκτωρα Μπόντεβικ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κριστόφσον Μπόντεβικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτη παρατήρηση, πρωτού ξεκινήσω την σύντομη ομιλία μου. Όταν μας ζητήθηκε να συντάξουμε αυτό το πρώτο έγγραφο, ε, αυτό έγινε πολύ πριν ο κύριος Γιούνκερ εξηγήσει το σχέδιο του και η επικέντρωσή μας ε, ε, επικεντρωθήκαμε στο πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα χρήματα του ΣΥΕΦ e και αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να εξετάσουμε τους διαδρόμους ε, και να, τις συζητήσεις που έχουν γίνει με πολιτικούς και εμπλεκόμενους φορείς. Και κατά τη συζήτησή μας με τους υπουργούς για τους διαδρόμους αναγνωρίστηκε ευρέως ότι οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν ε, σημαντικό στοιχείο για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Υπάρχει έλλειψη επενδύσεων στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρόβλημα, το πραγματικό. Είναι πρόβλημα και για το παρόν και για το μέλλον. Διότι αν η ε, έλλειψη επενδύσεων συνεχιστεί θα, θα υπάρξουν πολλά προβλήματα θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα γιατί θα υπάρξουν ανάγκες όσον αφορά την, ε, συν... τη συντήρηση και όλα αυτά θα δημιουργήσουν συμφόρηση στις υποδομές. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του Δούνου του επιβεβαιώθηκε ότι σήμερα θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στις υποδομές, ιδιαίτερα σε χώρους με χαμηλό ποσοστό ανάπτυξης και υψηλή ανεργία. Και ε, οι αυξημένες δημόσιες επενδύσεις είναι ε, ε, ένα από τα τελευταία εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας για την αύξηση της, για την ενίσχυση της ανάπτυξης και πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, βελτιώσουν τις δημόσιες, τα δημόσια οικονομικά τους και με πολλαπλασιαστικό ε, παράγοντα μέσω της συνεργασίας με οικονομικούς φορείς αλλά και με, μέσω της εξοικονόμησης κόστου συντήρησης και επισκευών που θα προκύψουν στο μέλλον και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της Eurostat που σήμερα δεν περιλαμβάνουν ένα τέτοιο κανόνα. Επίσης αναφέρεται ότι έως το 2030 θα χρειαστούν 1,5 τρισεκατομμύριο ε, σε επενδύσεις, ε, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών. Χρειαζόμαστε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι περιορισμένοι δημόσιοι πόροι κατανέμονται με τον ιδανικότερο δυνατό τρόπο. Και θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να συγχωνευτούν ε, τα ταμεία παρά να υποκαθιστούν το ένα το άλλο. Και σε αυτήν την, ε, από αυτή την άποψη είναι σαφές ότι υπάρχει ε, ζήτηση και θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτήν. Έχουμε ε, προσδιορίσει ανάγκης επενδύσεων ύψους 600 δισεκατομμυρίων για, τα, για το δίκτυο TNT. Από αυτά, τα 600 δισεκατομμύρια, ο συνάδελφός μου, ο κ. Κριστόφερσον, ε, προσδιορίσαν 127 δισεκατομμύρια ε, σε έργα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι κατάλληλα για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά ε, εργαλεία τα επόμενα χρόνια. Θα σας εξηγήσει ο κύριος Σέκη ε, αναλυτικότερα τι εννοώ με αυτό. Πώς θα καλύψουμε αυτές τις επενδυτικές ανάγκες. Είναι σημαντικό να συνδυαστούν διάφορες πηγές χρηματοδότησης από τις επιχορογήσεις, ε, την δημόσια χρηματοδότηση, αλλά βεβαίως και τις ε, επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Και είναι σημαντικό να μπουν στην συνολική εικόνα, να μπουν στο παιχνίδι και ιδιώτες επενδυτές για να αξιοποιηθούν τα 600 δισεκατομμύρια του CEF, για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες των 600 δισεκατομμύρων. Συγκεκριμένα, ε, ε, μακροπρόθεσμοι επενδυτές όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες ε, θα πρέπει να ε, απολαμβάνουν κατάλληλων προϋποθέσεων και με αυτό να περάσω στην επόμενη ε, διαφάνεια για το πώς μπορεί να ενισχυθεί, να ενεργοποιηθεί η ε, να ενεργοποιηθούν οι ιδιωτικές ε, επενδύσεις. Χρειάζεται σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, ένας αγωγός έργων. Χρειάζεται ε, μια μακροπρόθεσμη ορατότητα των έργων προκειμένου να προσελκυστούν ιδιώτες επενδυτές. Χρειαζόμαστε τεχνική αρρωγή, στεναρή από τα κράτη-μέλη για το πώς θα μπορέσουν να προσελκύσουν ιδιώτες ε, επενδύσεις και πώς θα μπορέσουν να δημιουργήσουν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού ταμείου. Αυτό μπορεί να γίνει και με την εξωτερική υποστήριξη, όπως για παράδειγμα από τις αναπτυξιακές τράπεζες ή από τις ε, κατάλληλες ομάδες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και με την δημιουργία ε, κοινών έργων και με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Είναι επίσης σημαντικό να προβλέπεται και να υπάρχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο. Η χρήση των χρηματοδοτικών συστημάτων προϋποθέτει απλουστευμένες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ε, ε, σταθερό επενδυτικό περιβάλλον το, το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να είναι σαφέ. Όσον αφορά τι κρατικέ επιχορηγήσεις θα πρέπει επίσης να υπάρχουν σαφείς κανόνες και διαδικασίε ελέγχου. Κάποιες ε, θα πρέπει επίσης να ε, προβλέπονται και συγκεκριμένε ομάδες έργων. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ε, προτεραιότητα ορισμένων έργων έναντι άλλων. Οι δημόσιες εγγυήσεις είναι άλλος ένας πυλώνας που μπορούν να ε, κινητοποιήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Και από αυτή την άποψη οι ευρωπαϊκές ε, εγγυήσεις, όπως αυτές που, στις οποίες προβαίνει η ΕΤΕΠ, θα πρέπει να διευρυνθούν. Τέλος, γνωρίζετε όλοι ότι οι υποδομές μεταφορών αποφέρουν κέρδη οικονομικά και κοινωνικά που πολλές φορές δεν αποτιμούνται σε χρήματα. Για παράδειγμα, η αρχή του ρηπαίνοντος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να διευρυνθεί περισσότερα ώστε να ελαφρυνθούν οι φορολογούμενοι. Και κατά τη γνώμη μου η χρήση οικονομικών δομών, χρηματοδοτικών δομών που σχετίζεται με την ε, ε, απόσταση είναι ο καλύτερος τρόπος να ε, βοηθηθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Schemes between the different modes of transport. Επίσης μπορούμε να έχουμε λίγο διαφορετικά οικονομικά ε, προγράμματα ανάλογα με, τους, με τα διάφορα είδη των μεταφορών. Επίσης μπορούμε να δούμε πώς ε, η οικονομική προσφορά μπορεί να ενισχυθεί. Ο... Ε, θα ήθελα επίσης να πω ότι θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτηση για τα ρυθμιστικά ζητήματα, τα οποία ε, πρέπει να εξεταστούν, όπως για παράδειγμα η περίπλοκη διαδικασία αδειοδότησης και δημοσίων προμηθειών, πρέπει να υπάρχουν απλούστεροι εναρμονισμένοι κανόνες σε σχέση με τα διάφορα ε, στάδια κατασκευής, ε, όλοι οι παράγοντες κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ενδεχομένως για καθυστέρηση στην κατασκευή ε, πρέπει να, να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Και όπως είπα και προηγουμένως ε, πρέπει να έχουμε καλύτερους ε, κανόνες κρατικούς και πρέπει να δούμε επίσης και τα στατιστικά στοιχεία ε, των ε, διαδικασιών. Η φερεγγιότητα επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να συζητήσουμε για αυτό το θέμα μετά την παρουσίασή μας. Ένας τρόπος ακόμη ενίσχυσης των οικονομικών προσφορών είναι να υπάρχει μια προσέγγιση κύκλου ζωής συμπεριλαμβάνει στο κόστος όχι μόνο την κατασκευή αλλά και τη συντήρηση και τη λειτουργία βλέποντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής και μόνο τότε μπορεί να υπάρχει βιωσιμότητα στο πρόγραμμα, ε, ε, να είναι επιχειρησιακό το πρόγραμμα και επίσης να μην υπάρχουν ε, προβλήματα με την ζημιές με την χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σέκη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για ε, την ε, πρόσκληση. Θα ήθελα να συνεχίσω χωρίς να επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν ήδη, αλλά θα προσπαθήσω να εμβαθύνω σε μερικά άλλα σημεία της κοινή δουλειά μας. Βλέπετε εδώ έναν πίνακα, ο οποίος δίνει ένα παράδειγμα των τομέων που είναι επιλέξιμα για τα νέα οικονομικά προγράμματα. Και τι εννοούμε με αυτό, θέλαμε να παρουσιάσουμε αυτόν τον κατάλογο όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με καινοτόμο χρηματοδότηση, στι ε, στις περισσότερες περιπτώσεις δηλαδή ένα συνδυασμό ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ε, η προσέγγιση συγχώνευσης για να το πούμε έτσι στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Εδώ είναι ενδιαφέρον ο κατάλογος γιατί έχουμε 127 δισεκατομμύρια που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς και πρέπει να προσθεθεί στον κατάλογο αυτών τα συστήματα διαχείρισης της ε, κυκλοφορίας όπως το RTMS, ε, το CESAR, το RIS, το ITS κλπ. Όπως επίσης ε, κάποιους ε, στόλους που πρέπει να προσαρμοστούν ε, σε συστήματα ε, καθαρότερα, όπως επίσης και την ανάπτυξη υποδομή για καθαρά καύσιμα. Εκτός από αυτά βέβαια υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό επενδύσεων Μπορεί να σας κάνει εντύπωση ο αριθμός, το ποσό που έχει να κάνει με τις σιδηροδρομικές και στις μεταφορές, 29 δισεκατομμύρια, αλλά είναι ένα τμήμα του συνολικού ποσού που έχει να κάνει ε, σε, με, μικρότερες, ε, με μικρότερο σιδηροδρομικό δίκτυο που έχει να κάνει με τη μεταφορά στο αεροδρόμιο από και προς, είναι ε, άλλα, άλλοι τομείς που είναι πιο περίπλοκο να χρηματοδοτηθούν. Μπορούμε όμως να φανταστούμε ότι θα, υπάρξει, θα υπάρξουν τμήματα στη χρηματοδότηση, όπως για παράδειγμα μπορούμε να φανταστούμε το ERTMS, που θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για έναν ιδιωτικό, ιδιώτη επενδυτή. Οπότε ζήτηση υπάρχει και ε, εξακολουθούμε να προσπαθούμε να εντοπίζουμε προγράμματα ε, που είναι κατάλληλα και ε, βάση του προγράμματος Juncker. Τι συμβαίνει τώρα. Μια κοινή εργασία από τους συντονιστές των διαφόρων διαδρόμων, του ERTMS, του, των αυτοκινητοδρόμων, Επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προετοιμάζει τις επενδύσεις για το πρόγραμμα ε, ε, Juncker και επίσης πρέπει να εντοπιστούν ορισμένα προγράμματα σε κάθε διάδρομο για να υπάρχει κάτι έτοιμο προς χρηματοδότηση αν όλα πάνε κατευχήν. Έχει ήδη αναφερθεί ότι Αφού θα έχουμε εντοπίσει όλα τα κατάλληλα για χρηματοδότηση προγράμματα θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την έκθεση μέχρι το 2015 το μήνα Ιούνιο και θα γίνουν συναντήσεις όχι μόνο με την ΕΤΕΠ, κάτι που έχει ήδη προβλεφθεί, αλλά και με τα, τις αρχές των κρατών μελών προκειμένου να ε, ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις και σχόλια. Επίσης ε, ε, ε, θα συνεχιστούν θα συνοχιστούν εργασίες που θα συνοδεύσουν τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσον αφορά τα προγράμματα χρηματοδότησης για τις ήπιες υποδομές που θεωρούμε ότι είναι πολύ, πολύ κατάλληλα και ε, παρουσιάζουν ιδιαίτερο δυναμικό. Έχουμε επίσης ε, ένα διαρθρωμένο διάλογο με τους επενδυτές. Δεν χρειάζεται να αναφέρω όλα αυτά που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια γιατί αναφέρθηκαν προηγουμένως. Τώρα, το θέμα ε, των κινδύνων που πρέπει να καλυφθούν, τι θα θέλαμε να συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα και τι θα θέλαμε να χρηματοδοτηθεί και ποιο είναι το καλύτερο οικονομικό μοντέλο που ε, έχουμε στη διάθεσή μας. Ακόμη πιο σημαντικό και από τη διαβούλευση με τους ε, πιθανούς επενδυτές, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ε, ως προς την αναγνώριση των εμποδίων και των πιθανών λύσεων. Υπόθηκε και προηγουμένως από τους συναδέλφους, αλλά θα το ξαναπώ. Αυτή η δουλειά που έχει γίνει από τους ε, υπουργούς μεταφορών μας ε, είχε ξεκινήσει ήδη από το πρόγραμμα, πριν από το πρόγραμμα Juncker και σκοπό είχε να εξεύρει τρόπους να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη χρηματοδότηση μέσω της, οικονομικής, ε, της χρηματοδοτικής καινοτομίας θα θυμάστε ότι παλιά μιλούσαμε για project bonds και τέτοιου είδους ε, μέσα. Συνεχίζουμε λοιπόν την εργασία μας προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με ιδιωτικούς επενδυτές γιατί ε, οι διαδικασίες αυτές, οι PPP ήταν υπόψη, τις είχαμε υπόψη μας ήδη πριν από, ε, από το πρόγραμμα Juncker και ειδικότερα σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη που εξακολουθούν να ε, θεωρούνται ως καλύτερες πρακτικές. Λοιπόν, καινοτομία για τη χρηματοδότηση λοιπόν, εμπόδια, ρυθμιστικό πλαίσιο, όλα αυτά ε, δημιουργούν πρόβλημα ε, στη σχέση προσφοράς και ζήτησης. Αυτό είναι το σημαντικότερο τμήμα της δουλειάς μας, γιατί όλα αυτά τα εμπόδια κανονικά προέρχονται αποφάσεις που λαμβάνονται από κάποιον και ε, από κάποιο φορέα και εφαρμόζονται από κάποιον άλλο φορέα ε, ο οποίος προφανώς ζηλεύει τα προνομιά του είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει κανείς κάποιον τέτοιο φορέα να αλλάξει γνώμη. Και πάση περιπτώσει δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να εντοπίσουμε τα εμπόδια, να προτείνουμε πιθανές λύσεις, και μετά να το αφήσουμε σε εκείνους που έχουν την ευθύνη να ε, λάβουν την απόφαση. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό και είναι ο λόγος για τον οποίο ολοκληρώνοντας ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας ε, στην δουλειά μας γιατί νομίζω ότι πάρα πολύ χρήσιμες προτάσεις ε, και σχόλια μπορούν να προκύψουν και από εσά. Ευχαρίστως να τις λάβουμε υπόψη και να τις ενσωματώσουμε. Και βεβαίως ε, δεδομένη της πολιτικής σας ευθύνης, ελπίζουμε ότι γνωρίζετε τι διακυβεύεται και αν θεωρείτε ότι είναι κάτι καλό αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, παρακαλούμε υποστηρίξτε μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτές τις τρεις παρουσιάσεις είχαμε. Ανοίγει ο κατάλογος ομιλητών. Πρώτος ο κύριος Βιρβαντεκάμπ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όσο, όσον αφορά το θέμα θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις κυρίους. Πολύτιμη ήταν η παρουσίαση των πληροφοριών που έκαναν. Τους ευχαριστούμε και για την έκθεση και ευχαριστούμε και για την προφορική παρουσίαση. Προφανώς βρισκόμαστε μεταξύ συμπληγάδων πετρών εδώ. Έχουμε την έκθεση και από την άλλη πλευρά τα καθημερινά θέματα που συζητούμε. Η κυρία Γιάλα Σέντερ η ε, συνάδελφος θα αναφερθεί σε αυτό. Ε, όταν διάβασα την έκθεση θεώρησα ότι ήρθε πολύ αργά. Βλέποντας την έκθεση και διαβάζοντας προσεκτικά μπορεί να μάθει κανείς πολλά. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε και αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα κριτήρια, ποια θα είναι η βάση ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εγκρίνει τα διάφορα έργα. Έχουμε τα διάφορα έργα που προβλέπονται στο ΣΕΦ, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τούτων λεχθέντων έχω κάποιες ερωτήσεις. Οι συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα δεν έχουν αποδείξει ότι αξίζουν ακόμα. Κοστίζουν πολλές μεγάλες προσπάθειες για να ε, υλοποιηθούν σωστά και να είναι επιτυχείς και αν μπορούσε κανείς να ετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές, να ετοιμάσει ένα εγχειρίδιο για τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, αυτό θα ήταν χρήσιμο. Για την ώρα η όλη προσπάθεια είναι πολύ χρονοβόρα. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Δεύτερον, οι συνδυασμοί των διαφόρων ε, διάβλων χρηματοδοτήσεως. Έχουμε επιδοτήσεις από το ΣΕΦ, έχουμε δάνεια, που χορηγούνται και μετά και ιδιωτικού πόρους. Και αυτή η ανάμιξη δημιουργεί δυνατότητες αλλά είναι πολύ τεχνικά περίπλοκο να λειτουργήσει όλο αυτό. Τρίτο θέμα. Πώς μπορούμε τα ιδιωτικά χρήματα, τα χρήματα των ιδιωτών να τα έχουμε στη διάθεσή μας. Ας δούμε τις γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες. Διαθέτουν πολλά χρήματα. Πώς θα απελευθερωθούν οι πόροι όμως. Έχουμε κανόνες περιφερεγκαιότητας, αλλά η απόσβεση των επενδύσεων είναι μια άλλη πτυχή. Και σε μια τελική έκθεση θα ήθελα να δω περισσότερες λεπτομέρειες, κάποιες συμβουλές, το πώς τα ιδιωτικά χρήματα θα μπορούσαν να επενδυθούν για έργα δημοσίων υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι άλλο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ήδη μιλήσατε με αυτήν. Η τελική σας έκθεση θα ολοκληρωθεί αρκετά έγκαιρα διότι ξέρω ότι λαμβάνονται πολλές πολιτικές αποφάσεις σε αυτή τη συγκυρία. Είπατε θα προσπαθήσετε να τελειώσετε μέχρι τον Ιούνιο. Μήπως διατέχετε κάποιο κίνδυνο, μήπως είναι επικίνδυνη αυτή η κατάσταση. Σας το θέτω σαν ζήτημα. Ευχαριστώ. Ισμαήλ του έχει το λόγο. Ευχαριστώ. εκ μέρους της ομάδας των σοσιαλιστών για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση της έκθεσης και από τους τρεις ομιλητές, τους τρεις συναδέλφους. Είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και κάποιες εβδομάδες από τότε που η Κομισιόν Juncker πρότεινε αυτό το EFSI και φυσικά ως Επιτροπή Μεταφορών προβληματιζόμαστε κατά πόσο τα διάφορα κριτήρια που είχαμε θεσπίσει στο CEF και, στο, και στις κατευθυντήριες γραμμές για το TNT θα χρησιμοποιηθούν και κατά την επιλογή των έργων αν δηλαδή θα ε, χρησιμοποιηθούν τα ίδια κριτήρια κατά την επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν. Να σημειώσω επίσης ότι τις τελευταίες εβδομάδες με την Γενική Διεύθυνση MOVE και με την Επιτροπή έχουμε συζητήσει και μάθαμε τελικά πώς τελικά θα προκύψουν αυτά τα 315 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει κανείς που δεν τα θέλει, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε σε κάθε περίπτωση ότι ε, στην πραγματικότητα τα πραγματικά χρήματα είναι 8 δις. Είναι τα 3,3 από το ΣΕΦ, από το, τα 2,7 από το ορίζοντας 2020 και 2 δισεκατομμύρια από μη αξιοποιημένους πόρους του προϋπολογισμού. Ε, που συνολικά μας κάνουν 8 δις ε, και άλλα 8 δις που βάζει το, το ταμείο αυτό. Άρα συνολικά 16 δισεκατομμύρια και με αυτά ε, πρόκειται να εξευρεθούν 315 δισεκατομμύρια. Και 315 να μην είναι και να τελικά να αποτελέσουν μόνο, να φτάσουμε μόνο στα 100 δις, πάλι επιτυχία θα είναι. Αν δούμε τα έργα που έχουν ε, προταθεί μέχρι στιγμής, θα δούμε ότι το 29% αφορού, αφορά το, τον τομέα των μεταφορών και αυτό δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα. Νομίζω ότι το, σημαντικότερο ερώτημα το έχετε θίξει κι εσείς με την έκθεσή σας. Δηλαδή, ποια είναι τα εμπόδια τελικά. Σε τελική ανάλυση σκοπός είναι να παρακινήσουμε ιδιώτες επενδυτές να κάνουν επενδύσεις. Άρα ποια είναι τα εμπόδια που υπήρχαν μέχρι τώρα. Για παράδειγμα χρειάζεται μήπως ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα, τους, ε, που θα παρέχει βοήθεια σε εκείνους που θα βάλουν τα χρήματα στην πραγματικότητα. Υπήρχε και παλαιότερα ένα τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο, υπάρχει ακόμη, αλλά θα πρέπει η Κομισιόν να σκεφτεί μήπως ε, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου ε, ε, μήπως αυτή τη φορά θα πρέπει να αποτραπεί ένας ανταγωνισμός μεταξύ των ε, γενικών διευθύνσεων και έτσι θα κερδιθούν επενδυτές. Αναφερθήκατε και σε ένα άλλο θέμα. Τα έργα υποδομής που θα χρηματοδοτηθούν από αυτό το ταμείο, αν θα πρέπει να ε, ε συνάδουν με τα κριτήρια του, του Μάστριχτ αν θα συνυπολογίζονται. Ε, και ακούσαμε για πρώτη φορά ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβαίνει, ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη, αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Επίσης υπάρχει μια τεχνική αρρωγή όσον αφορά τις ε, τεχνικές άδειες κτλ. Επίσης πολύ θετικό. Κάτι που μου άρεσε και θέλω να το πω είναι αυτή η προσέγγιση κύκλου ζωής. για μένα είναι, είναι μια εξαιρετική ιδέα. Γιατί αυτή ήταν και η δική μας προσέγγιση στα νομοθετήματα που έχουμε ε, θεσπίσει. Γιατί υπήρξαν και έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν χωρίς να έχει, να έχει ληφθεί υπόψη το μέλλον, ποια θα είναι τα μελλοντικά κόστη δηλαδή. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ε, πάντοτε να εξετάζουμε και τις παράπλευ, τα παράπλευρα κόστη, για παράδειγμα το οικολογικό αποτύπωμα, το αποτύπωμα άνθρακα, για να μπορεί να γίνεται μια συνολική αξιολόγηση κάθε έργου. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να ε, συμπεριληφθεί ε, και στην ομοθεσία που θα δημοσιευθεί, το λέω και στους δύο συνεισηγητές μας, και τέλος Όσον αφορά αυτήν την, αυτήν την, αυτό το, τη μόχλευση που θέλουμε να επιτύχουμε. Αν, θέλω να θέσω το ερώτημα, αν αυτή η μόχλευση είναι ρεαλιστική. Υπάρχουν και μελέτες, για παράδειγμα του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πράγματα μάλλον δεν δημιουργούν τόσο μεγάλη αισιοδοξία όσον αφορά την κερδοφορία ε, των ε, επενδύσεων. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Εν πάση περιπτώσει η συζήτηση θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ ο Ρόμπερτ Ζήλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Όπως γνωρίζετε, στην Επιτροπή μας ε, μας απασχολεί κάπως ε, η εφαρμογή του προγράμματος και ειδικότερα για την πολιτική μεταφορών ε, και ειδικότερα για τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τα προγράμματα των διαδρόμων και τη διαχείριση των διαδρόμων. Έχετε πολύ πείρα σε αυτό και το είδα και από την παρουσίασή σας νομίζω ότι ελπίζω ότι θα μπορέσετε να μας δώσετε κάποια απάντηση σε σχέση με το πρόγραμμα Juncker, τέλος πάντων κάποια πιο αισιόδοξη θεώρηση. Έχω τις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, αυτούς τους διαδρόμους πώς τους βλέπετε, για ποιο λόγο να επιλέξουν οι ιδιώτες επενδυτές κάτι τέτοιο αντί των αυτοκινητοδρόμων. Ίσως η DigiMove μπορείτε, μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα τις επιδοτήσεις που αφορούν τις διευκολύνσεις στους διαδρόμους. Αν η DigiMove μπορεί να μπλακεί κάπως περισσότερο στην επιλογή ε, των προγραμμάτων, να συμμετέχει στην Επιτροπή Επιλογής των Προγραμμάτων, αν η DigiMove κρατήσει τις επιδοτήσεις για τους διαδρόμους, σε αυτή την περίπτωση ίσως να προτιμηθούν οι διάδρομοι αυτοί και από τους ιδιώτες. Όμως υπάρχει μια αμφιβολία λόγω του προγράμματος Juncker γιατί μπορεί αυτά τα προγράμματα να διαρκέσουν 10-15 χρόνια και είναι εντελώς διαφορετικό το χρονικό όριο. Οι ιδιώτες ε, επενδυτές ε, θέλουν κάποια απόδοση για την επένδυσή τους μετά από 3-4 χρόνια. Έχουμε και κάποιες ε, περιοχές με ε, προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης ε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις περιοχές να γίνουν υποδομές. Πώς μπορείτε, ότι Πώς μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα Juncker να βοηθά αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν βλέπω ε, από πού μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες και από οικονομικής απόψεως. Εσείς κύριε Κριστόφερσεν είπατε στα εισαγωγικά σας σχόλια ότι η σημασία του προγράμματος Juncker και ειδικότερα για τις επενδύσεις στις μεταφορές είναι αύξηση της απασχόλησης. Πάρουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε επενδύσεις ε, από ασφαλιστικά και συνταξιδοτικά ταμεία από την κυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια έχει φύγει, έχει ε, έχει αντικατασταθεί ε, από χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το EFSI κλπ. Για ποιο λόγο λοιπόν ε, να ε, τα χρήματα αυτά από το πρόγραμμα Juncker να πάνε στην Ελλάδα ε, εφόσον πριν από δύο χρόνια που υπήρχαν, υπήρχε αυτή η χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση αυτή τελικά αφαιρέθηκε από την Ελλάδα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Το θέμα της για τα διόδια όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα Juncker. Δεν δημιουργείται καμία ε, ισορροπία αν δεν είναι πραγματικά διόδια, αλλά είναι μια επιστροφή ε, επενδύσεων, μια απόδοση επενδύσεων μετά από 30-40 χρόνια ε, μιας ε, επένδυσης. Αυτά τα χρήματα πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ένα συγκεκριμένο οικονομικό έτος το 2016 για παράδειγμα που μπορεί να τρέχει ένα πρόγραμμα. Αν αυτή η χώρα θα πρέπει τα χρήματα αυτά να τα βάλει στον ισολογισμό του για 20 χρόνια. Υπάρχει και το Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξη. Νομίζω ότι σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Juncker μπορεί μετά να επέλθει καταστροφή. Και μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και του τρει ε, ομιλητέ Σύντομα, θα τα πω γιατί πρέπει να φύγω σε μια άλλη επιτροπή για την μια ψηφοφορία οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να, να περιμένω καν ε, να ακούσω τις απαντήσεις αλλά θα με ενημερώσουν ε, οι βοηθοί μου ε, και ε, φαντάζομαι ότι και οι συνεισηγητές μας η κυρία Μπιλμπάου και ο κύριος Ρικέ θα θέσουν και εκείνοι ορισμένα ερωτήματα. Φυσικά ακούγεται τέλεια. Ε, τέλειο να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και το Connecting Europe Facility για τους διαδρόμους και το σχέδιο Juncker. Φυσικά μας φαίνεται μάλλον ε, άσχημα το γεγονός ότι αφαιρούνται χρήματα από, το, από τις μεταφορές και μετακυλίονται σε άλλους ε, κλάδους. Εγώ προσωπικά δεν είμαι τόσο αρνητική γιατί θεωρώ ότι και οι δρόμοι αποτελούν ε, τμήμα των διαδρόμων και οι γέφυρε, για παράδειγμα, ε, οπότε είναι θετικό το να προσελκυστούν ιδιωτικέ επενδύσεις. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Τις εξή. Είπατε ότι 100, έργα αξίας 127 δισεκατομμυρίων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ιδιωτικά κεφάλαια, δηλαδή επενδυτές ιδιώτες, Το ερώτημά μου είναι υπάρχει κάποια περιφερειακή κατανομή αυτών των ε, χρημάτων και δεύτερον σε ποιο βαθμό τα έργα που θεωρούνται χρήσιμα ε, Κατά πόσο λοιπόν αυτά τα έργα θα έχουν μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη εξία, ένα κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε και στο CEF όπου είχαμε πει ότι θα πρέπει να είναι χρήσιμα τα έργα και θα πρέπει με κάποιον τρόπο να φέρουν και ένα πλεονέκτημα, μια προστιθέμενη αξία δηλαδή για τους πολίτες και τους καταναλωτές. Οπότε φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα συμβαίνει, θα ισχύει, αλλά σε ποιο βαθμό βλέπετε εσείς να ε, ανταποκρίνετε στην πραγματικότητα αυτή η επόθεση που κάνω για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη ε, αξία. Και μια τελευταία παρατήρηση, είπατε, δηλαδή, είπατε για το earmarking, δηλαδή για τον ε, διορισμό συγκεκριμένων στόχων, όπως για παράδειγμα ε, με τους ε, δρόμους με διόδια. Ξέρετε ότι στη Γερμανία υπάρχει μια σχετική συζήτηση και αν τελικά αποφασιστεί ότι κάτι, ότι μπορεί να γίνει, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει στη Γερμανία, αλλά μόνο εφόσον υπάρχουν και συγκεκριμένες ε, δεσμεύσεις. Ίσως είναι και αυτός ένας τρόπος για να προσελκυστούν χρήματα στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Το, ε, η αρχή user base ε, ο χρήστης πληρώνει, ε, είναι χρήσιμο. Ε, υπόθηκε όμως ότι, το, ότι ο ξένος, ο πληρώνουν οι ξένοι δεν είναι σωστή προσέγγιση. Η κυρία Ντελή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας ως εμπειρογνωμόνων, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για τις συγκεκριμένες ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση μέσω μέσων, είτε με συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα ή τα project bonds. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο μου ερώτημα είναι πώς και πότε τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, λάβουν αυτή τη δανειοδότηση για την εφαρμογή προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Juncker. Επίσης, πόσες βιώσιμες θέσεις απασχόλησης σήμερα μπορείτε να υπολογίσετε όταν χρηματοδοτείτε ένα πρόγραμμα, ειδικότερα όταν είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για ένα μεγάλο ε, πρόγραμμα που είναι το ε, Λιόν Τωρίνο νομίζω ότι σήμερα από απόψε ως αντικτύπου έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία να μας πείτε και να μας πείτε βάσει αυτών των στοιχείων πρέπει να, να επενδύσουμε σε αυτό το είδος προγράμματος γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρη γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει η ε, χρηματοδότηση και δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη έχουν τέτοιου είδους ε, πόρους. Ευχαριστώ η κυρία Ίνες Αγιάλα Σέντερ, έχει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ Προέδρε, συγγνώμη για τη φωνή μου. Ελπίζω να μπορέσω να ολοκληρώσω χωρίς να χάσω τη φωνή μου. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες. Έχω κάποιες ερωτήσεις και για τους τρεις. Καταρχάς προς τον κύριο Κριστόφερσον θα ήθελα να σας ρωτήσω επειδή ξέρετε στις βάθος το σύστημα τη ε, της διαχείρισης των διαφόρων ε, ταμείων και λοιπόν και τη διάθεση των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ε, είχατε τη δυνατότητα να εκτιμήσετε πόσα χρήματα υπάρχουν και προβλέπονται στον ευρωπαϊκό προπολογισμό για τους σκοπούς αυτούς. Πέραν των όσων ε, βρίσκονται στο ΣΕΦ για επενδύσεις στις υποδομές. Θα χρειαστούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα πρέπει να συμπληρώσουμε τόσο διατίθεται από το ΣΕΦ και να προσαρμόσουμε αναλόγως τα επενδυτικά πακέτα. Καμιά φορά ίσως να μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από, τα, από θεματικό, από μη χρησιμοποιημένα κονδύλια. Αλλά αυτό που δεν θα πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε χρήματα από τα κονδύλια του ΣΕΦ. Γιατί δεν διαθέτει και τεράστιους πόρους. Πρώτα απ' όλα αναφερθήκατε σε φραγμούς που αποκαρδιώνουν τους ιδιωτικούς ε, επενδυτέ. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό, δεν ξέρω λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, διότι επί παραδείγματι κατά το παρελθόν εξετάσαμε το θέμα των κρατικών ενισχύσεων όταν μιλούσαμε για την Νότια ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήθηκε μεγαλύτερη ευελιξία. Και νομίζω ότι είναι ανησυχητικό αυτό που αναφέρεται. Χτυπάει το κουδούνι του συναγερμού διότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το θέμα αυτό. Σε κάποιες χώρες χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις και μεγαλύτερη ευελιξία εκεί θα ήταν καλή αν είχαν πλεόνασμα στους προπολογισμού τους. Διαφορετικά δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Τίθεται και το θέμα του αντικτύπου για το περιβάλλον. Είναι κάτι που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε αξιολόγηση έργου. Όσον αφορά τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά μέσα, Έχουμε δύο εκδοχές, έχουμε το ΣΕΦ και εντός αυτού έχουμε μακροχρόνια χρηματοδότηση και άλλα είδη χρηματοδοτήσεως. Άρα έχουμε χρηματοδότηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη συνταξιδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείε που θα ενδιαφερόταν να επενδύσουν σε αυτού του είδους τα έργα για υποδομές των μεταφορών και πρόσφατα στα πλαίσια του πακέτου Juncker τονίστηκαν οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και οι επενδύσεις αλλοδαπών όπως είναι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Ε, ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ όλους σας για τις παρουσιάσεις σας. Ήταν άκρος ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά που έθιξα. Και ποια είναι η άποψή σας, πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει το κάθε εργαλείο. Ποιο είναι το μέγιστο που μπορούμε να πετύχουμε με το ΣΕΦ και πώς, όσον αφορά συγκεκριμένα έργα. Πώς μπορούμε να πετύχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατό Λοιπόν, όσον αφορά τις επενδύσεις πρέπει να συζητήσουμε και τι γίνεται όσον αφορά τα θέματα τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που είπατε Αναφερθήκατε στη δυνατότητα να μην εφαρμοστεί, ή να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο, να εφαρμοστούν διαφορετικά οι κανόνες ε, του Μάστριχτ. Κυρίως αναφερθήκατε σε διάφορες δυσκολίες που εμποδίζουν τις επενδύσεις. Θα ήθελα να γνωρίζω ποιες είναι οι απόψεις σας. Κύριε Σέκη, ε, σας γνωρίζουμε όλοι. Είσαστε υπέρ της διασταυρούμενης χρηματοδοτήσεως. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε εκεί Παραδοσιακά είμαστε κατά. Όσον αφορά το Solvency 2 και τη Βασιλεία 3, ε, δύο πακέτα που έχουν εγκριθεί, ο στόχος εκεί ήταν να αποφευθεί κάθε τραπεζική καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα εργαλείο που ίσως να είναι καλό, αλλά ίσως πλέον ευαίσθητο. Έχουμε και τα ομόλογα έργου που μέχρι τώρα είχαν προταθεί και ε, νομίζω ότι απέτυχε αυτή η πρόταση. Όσον αφορά τη διαχείριση, τη διακυβέρνηση, πώς μπορούμε να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε ξανά τέτοιου είδου αποτυχίες. Dominique κρικέ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ τους τρεις ε, φιλοξενούμενους που παρενέβησαν για τη δουλειά τους. Εστιασμένοι, Βιάνα πέσανε. Και ξεκίνησαν ε, πριν να βρεθούμε στην όλη κατάσταση της αβεβαιότητας που είμαστε σήμερα. Να πω κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η σημασία των μη χρηματοστατικών εμποδίων. Η συζήτηση αφορά το σχέδιο Juncker, τα χρηματοστατικά ε, εργαλεία ορίζοντας 2020, το ΣΕΦ, συζητούμε τη χρηματοδότηση, αλλά υπάρχουν εμπόδια μη χρηματοδοτικά, μη χρηματοδοτικά. Η οριμότητα των έργων, η ποιότητα των έργων, το πρόβλημα της συντήρησης των υποδομών, ο κύκλος ζωής των υποδομών και τα ρυθμιστικά εμπόδια είναι ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να χάσουμε αυτά ε, τα σημεία όταν τα συζητάμε. τα εμπόδια τα ρυθμιστικά είναι σημαντικά και για τα έργα και για τη χρηματοδότηση. Τα αναφερθήκατε κατοικές ενισχύσεις, τα επιβαλλοντικά προβλήματα, οι δημόσιες προμήθειες, όλα αυτά που περιπλέκουν κατά σημαντικό τρόπο τη βιωσιμότητα ή την προβλεψιμότητα ενός έργου. Και από πλευρά χρηματοπιστωτική η ρυθμιστική ε, πτυχή, ε, βασιλεία 3, αφαιρεγκαιότητα 2 κλπ. Έχουμε έργα κοινοφελούς σημασίας. Εκεί δεν υπάρχει απόσβεση των επενδύσεων ή κέρδος και δεν μπορεί να γίνει συγχρηματοδότηση με ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν άλλα έργα αντιθέτω που ε, κάνουν απόσβεση των επενδύσεων και οδηγούν σε κέρδη που μπορεί να συμμετάσχει και ο ιδιωτικό τομέα και μεταξύ των δύο πρέπει να έχουμε κάποια έργα που είναι κοινοφελή αλλά αποσβαίνουν και τις επενδύσεις και πρέπει βρεθεί η σωστή ισορροπία. Να πληρώνει κανείς για το κοινοφελές ε, έργο ε, και τελικά να υπάρχει και ένα κέρδος που να καλύπτει τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα. Μπορούν να έχουμε θεμητές ανησυχίες. Θα ελπίζαμε ότι το πακέτο Juncker θα ε, ενίσχυε τις υφιστάμενες υποδομές, αλλά αντιθέτως μάλιστα θα τις αποδυναμώνει. Ε, πρέπει να κάνουμε και προτάσεις να μην κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση γιατί θα ήταν πάρα πολύ κακή αρχή για το σχέδιο Juncker. Κάποιες ερωτήσεις έχω, πρακτικής φύσεως. Αναφερθήκατε στην ομαδοποίηση των ε, ε, έργων διάβλος διοχέτευσης των έργων, αντιμετώπισης των έργων, συναρτήσει των τι αφορούν για να οριμάζουν με σωστό τρόπο. Να ομαδοποιούνται όταν είναι όριμα σε χαρτοφυλάκια. Ούτω ώστε να υπάρχει δυνατότητα ομαδοποίησης των επενδυτών. Δύο διαφορετικές ομαδοποίησεις. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε. Και για το pipeline αναφέρεται η πρόταση στα πλαίσια του ε, πακέτου Juncker αυτό πώς μπορούμε να περάσουμε από τη δρομολόγηση, από το διάβλο, από το pipeline στο χαρτοφυλάκιο, η πορτφόλιο. Δεύτερον, αναφερθήκατε στην ομαδοποίηση γύρω στα μεγάλα οριζόντια έργα διαφόρων εταίρων διαφορετικών. Τα εναλλακτικά καύσιμα μπορεί να διαφέρει τους παραγωγούς ενέργειας, τους διανομής καυσίμων, παραγωγούς οχημάτων ηλεκτρικών ή ε, οχημάτων με υδρογόνο, των αυτοκινητοβιομηχάνων και τις χώρες πώς ομαδοποιείται φορείς τόσο διαφορετικούς. Από τη στιγμή που έχουμε δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο ή μια διεύλο, πώς δημιουργούμε ομαδοποίηση των επενδυτών. Υπάρχει τρόπος. Νομίζω ότι είναι τρεις προσεγγίσεις που μπορούν να βοηθήσουν να λειτουργήσουν καλύτερα αυτές οι προσπάθειες. Πρώτη ερώτηση. Από χρηματοστητική πλευρά, τι ρύθμιση μπορούμε να προτείνουμε Αναφερθήκατε στο Solvency 2 στην έκθεσή σας. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν πραγματική πρόταση για να ε, κινητοποιήσουν περισσότερο τους ιδιωτικούς πόρους. Τέλος, μια ερώτηση Παύλα Σύσταση. Ποια είναι η άποψή σας για τη δημιουργία ενός, το, για το καθεστώς εν, ε, ενός ευρωπαϊκού ευρωπαϊκού έργου μακροπρόθεσμου, δηλαδή, πώς το λέω, το σχέδιο Juncker ή το ΣΕΦ ή κάποιο άλλο μέσο, θέτει μια ετικέτα σε ένα έργο, το επιλέγει σαν χρηματοδοτούμενο, δυνατό να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Αν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θεωρεί ότι είναι επιλέξιμο ένα έργο, θα το αναφέρει. Θα δώσει κάποια εγγύηση από το Ταμείο Εγγύησης Οικονομικά παίρνει μια ετικέτα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, μια σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό είναι το σχέδιο Juncker. Μπορούμε αυτή τη σφραγίδα ούτω ή πίν ε, να μπορούμε να τη χορηγούμε πιο εύκολα μέσω απλούστευση των διαδικασιών. Αν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό έργο κοινοφερέ για την Ευρώπη, όχι μόνο θα υπάρχει εγγύηση οικονομική αναγκαία, αν θα υπάρχει και ιδιαίτερο καθεστώ για αυτό το έργο ρυθμιστικό, που θα οδηγεί σε ρυθμιστικέ απλουστεύσει όπως αυτές που αφορούν το περιβάλλον ή άλλες στοιχές ή όσον αφορά τις οικονομικές διαδικασίες για ενδεχόμενη εξέβρεση ενδιαφερομένων εταίρων. Αν έχετε ένα έργο ευρωπαϊκό σημαίνει ότι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να επενδύσουν σε αυτό το έργο και κάνοντας το αυτό ε, μπορούν να θεωρούν ότι καλύπτονται από 2. Μπορεί να υπάρχει ευρωπαϊκό έργο που θα έχει και ρυθμιστική εγγύηση πέρα από την οικονομική εγγύηση που θα χορηγείται εύκολα. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μάλλον. Γέλνς Νίλσεν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Ισχύει το γεγονός ότι το σχέδιο Γιούγκερ ανακοινώθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό. Πολύ βέβαια είχαμε σκεφτεί πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό στην πράξη και μέχρι στιγμή δεν έχουμε καταφέρει να ακούσουμε πολλά επ' αυτού του θέματος. Είναι βεβαίως θετικό να εξασφαλίζονται και οι δυτικές επενδύσει μακροπρόθεσμα. Φυσικά οι επενδυτέ δεν θέλουν να διατρέξουν υπερβολικά υψηλό κίνδυνο, ούτε θέλουν αποδόσεις 20 και 25%. Αλλά νομίζω για παράδειγμα ότι τα συνταξιδοτικά ταμεία αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Γνώμη μου είναι ότι στη Σουηδία το 20% ίσως όλων των κεφαλαίων ε, επενδύονται σε κρατικά ομόλογα. Και αυτά δεν είναι κερδοφόρα. Ενώ σε αυτού του είδους τις επενδύσεις ε, θα χρειαστούν σε κάθε περίπτωση ε, αποδόσεις που θα είναι υψηλότερες από εκείνες των κρατικών ομολόγων. Τα συνταξιδοτικά ταμεία αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητά τους, τη δυνατότητα να παρέχουν συντάξεις. Αλλά υπάρχουν και διάφορα είδη τα ταμεία δημόσια, ιδιωτικά και υπάρχουν και μικτού χαρακτήρα συνταξιδοτικά ταμεία. Και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι παράδειγμα και ασφαλιστικέ εταιρείε. Θα ήθελα να μάθω από εσά αν θεωρείτε ε, ότι υπάρχουν εμπόδια για την προσέλκυση και τέτοιου είδους μεικτών ε, συνταξιδοτικών ταμείων όσον αφορά τις επενδύσεις και θα ήθελα να ακούσω κάτι για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ε, υπάρχουν εμπόδια δηλαδή για την πραγματοποίηση τέτοιου είδους επενδύσεων. Και επίσης υπάρχει η ιδέα να υπάρχει μια ενιαία θερίδα. Καλή ιδέα, αλλά κατά τον προγραμματισμό της διάθεσης των δημόσιων ε, κονδυλίων ε, εμπλέκονται και συμπεριλαμβάνονται και συμμετέχουν και οι τοπικές αρχές και ε, δεν θα πρέπει να εξισωθούν φυσικά οι τοπικές αρχές με τις εθνικές αρχές. Κάτι τέτοιο θα ήταν βλαπτικό για τη δημοκρατία. Η κυρία Μπιλμπάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους ε, εισηγητές. Θα ήθελα να πω ότι έχω την πεποίθηση ότι το πρόγραμμα Juncker ε, θα είναι επιτυχές. Ε, πιστεύω όμως ότι εδώ αυτό στο βήμα μιλάμε για τα ίδια πράγματα επανειλημμένα. Ε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και το λέμε και σε εκθέσεις μας ότι πρέπει να εξαλείψουμε όλους τους φραγμούς που υπάρχουν σε διάφορους τομείς της ε, οικονομίας. Θα πρέπει να έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις, αυτό θέλουν όλοι, σε όλη την οικονομία θέλει ο κόσμος να μπορεί να επενδύει και θέλει να γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Χρειαζόμαστε καλύτερες συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα, είναι αποφελές για τους επενδυτές και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε τεράστιες ευθύνες. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά που διακυβεύονται και πάντα αντιμετωπίζονται ίδιες δυσκολίες. Δηλαδή η έλλειψη βούληση από πλευρά των κρατών μελών να κάνουν εκείνα τα οποία συζητούσαμε επί μακρόν. Έχουμε πολλά εργαλεία, έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας και όλα αυτά είναι καλά και άγια, αλλά αυτό που δεν κάναμε ήταν να απαντήσουμε σε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θέλουν πράγματι να άρουν τα εμπόδια για να υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα τα εμπόδια που εντοπίσαμε, αν δεν πάρουμε καταφατική απάντηση, τα μισά που συζητούμε θα παραμείνουν νεκρό γράμμα. Ε, γιατί τα λέω αυτά. Διότι είναι άλλο παράδειγμα του που μπορούν να πάρουν στραβόδρομα τα πράγματα. Χθε μιλούσα με κάποιου εκπροσώπου του συνδρομικού τομέα. Εκπροσωπούνται περίπου 10 διαφορετικέ εταιρείε και έλεγαν όλοι τα ίδια πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια για τι επενδύσει και για την πρόσβαση στην ε, αγορά και αν θέλουμε να υπάρξουν επενδύσεις πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια. Είναι πολύ επαχθής η όλη διαδικασία. Βέβαια, αν μιλάμε για τον τομέα της ενέργειας, αν συναντήσει κανείς εκπροσώπους του ενεργειακού τομέα, το ίδιο μήνυμα θα δώσουν. Και αν πάμε να συνομιλήσουμε με εταιρείε που είναι υπεύθυνε για τον ψηφιακό τομέα, θα πούν τα ίδια πράγματα, την ίδια ιστορία θα πούν ξανά. Λοιπόν, πώς θα απαλλαγούμε από τα εμπόδια είναι εμπόδια που έχουμε εντοπίσει σε πάρα πολλές εκθέσεις μας. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να βρουν λύση αν υπάρξει πολιτική βούληση. Ρωτώ το απλό ερώτημα. Υπάρχει πολιτική βούληση στα κράτη-μέλη για την άρση των εμποδίων. Και δεν είπαμε τίποτα για το τέταρτο συνδυδρομικό πακέτο και δεν ξέρουμε καν αν θα δει το φως της ημέρας. Υποτίθεται ότι απλουστεύει τα πράγματα, διευκολύνει τις επενδύσεις, διευκολύνει τη ζωή των επενδυτών και δεν είδαμε μεγάλη πρόοδο ούτε εκεί. Λοιπόν υπάρχουν, έχουμε πολλές ιδέες για σταθερότητα της αγοράς, σταθερό πλαίσιο επενδύσεων, κρατικές ενισχύσεις κλπ. Η πραγματικότητα όμως δυστυχώς είναι εντελώς διαφορετική εκφράζουμε μεγάλες ε, επιθυμίες και ευχολόγια, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τα κράτη-μέλη θα βγάλουν αυτά τα εμπόδια. Έχουμε πάρα πολλά έργα, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Ε, καθορίσαμε κάποια έργα που έχουν προτεραιότητα για μας για την επόμενη δεκαετία αλλά μέχρι το 2014 δεν είχαμε υλοποιήσει κανένα από τα μεγάλα προγράμματά μας που υποτίθεται ότι έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί ήδη. Και τώρα έχουμε άλλη μια δεκαετία μπροστά μας για τα προγράμματα. Πρέπει να δούμε πόσο επικερδής είναι οι επενδύσεις και πολλά κράτη-μέλη δεν επεξεργάζονται σωστά την προσέγγιση. Δεν προσπαθούν να άρουν τα εμπόδια. Χρειάζεται η πολιτική βούληση για να γίνει αυτό, να υπάρξουν επενδύσεις, να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες που θέλουμε. Κάνατε έξοχη δουλειά. Αυτό δεν το αρνούμε που δεν είναι. Έξοχη δουλειά που κάνατε. Και ε, γνωρίζω ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα για σας. Γνωρίζω ότι εξετάσατε διάφορους τομείς, ότι λάβατε υπόψη συστάσεις και σας λέω ειλικρινά, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα Κάθε έκθεση που συζητούμε ζητούμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή να απαλλαγούμε από τους διάφορους φραγμούς που υπάρχουν, που μας επισημαίνουν οι διάφοροι τομείς και είναι τεράστια εμπόδια για τις επενδύσεις. Θα πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά και ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να αναλάβουν κάποιες δεσμεύσεις σε πολιτικό επίπεδο, να υπάρξει πολιτική βούληση των κρατών μελών. Διαφορετικά το ΣΕΦ και το πρόγραμμα Juncker και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η συμμετοχή της, όλα αυτά θα κρέμονται στον αέρα και θα αφισβητήθει η επιτυχία όλων των προσπαθειών. Ζορς Μπαχ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους για το εξαιρετικό έργο που έχουν επιτελέσει. Συμφωνώ και εγώ με την συνάδελφο Μπιλμπάου. για τα νέα έργα και στο πλαίσιο του TNT. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό, αλλά κύριε Κριστόφερσον το είπατε κι εσείς για την, ε, για την ε, ανανέωση και τη συντήρηση των υπαρχουσών υποδομών και στην έκθεσή σας ε, αναφέρατε και κάποια προβλήματα, κάποιες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η κυρία Μπιλμπάου αναφέρθηκε στο ERTMS, αναφερθήκατε στο ΣΕΖΑΡ, στον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό, την αεροπορία Και καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα με την συνάδελφο. Όλα αυτά είναι κατηγορίες προβλημάτων που συζητούμε τουλάχιστον εδώ και δέκα χρόνια και διαπιστώνουμε ότι τα στα κράτη-μέλη δεν υπάρχει πολιτική βούληση να επιληθούν και αυτό θα είναι τελικά το μεγάλο θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε, αυτό το ζήτημα της εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών και επενδυτών. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς με τα σημερινά δεδομένα θα μπορέσουμε να πείσουμε επενδυτές να επενδύσουν σε αυτούς τους τομείς γιατί και εκείνοι ξέρουν τι έχει προηγηθεί γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα αντικρώμενες απόψεις και δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόοδος το ερώτημά μου είναι από πού αντλείτε εσείς τελικά αυτή την αισιοδοξία σας. Τα είπατε, τα περιγράψατε όλα με μεγάλη σαφήνεια, ε, είπατε και πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα έργα, μακροπρόθεσμα, αλλά από πού αντλείτε εν τέλει εσείς την αισιοδοξία που εμείς τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό έχουμε χάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρος εγώ είμαι ο τελευταίος ομιλητής και μετά θα μας απαντήσετε. Το σχέδιο Juncker έχει τρεις στόχους. Το είπατε κι εσείς. Θέσεις απασχόλησης, διασύνδεση της Ευρώπης και υπάρχουν βεβαίω και οι στόχοι για το κλίμα. Και το θέμα τώρα είναι να επενδυθούν χρήματα σε αυτούς τους τρεις στόχους. Όλοι έχουμε εμπειρία και γι' αυτό ίσως ακουγόμαστε και κάπως απεσιόδοξοι. Θέλαμε να υπάρξει ευρωπαϊκή ενοποίηση και στο δίκτυο σιδηροδρόμων που μοιάζει με κουρελού και ακριβώς τα κενά είναι εκεί που υπάρχουν και τα τα, τα σύνορα. Ε, τα τελευταία 20 χρόνια έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια και παρόλα αυτά δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο. Και τώρα ε, λέμε ότι α, τώρα έχουμε ακόμα περισσότερα, ακόμα περισσότερα χρήματα. Α, ωραία, ας κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα έργα. Εκατό εκατομμύρια χρειάζονται για τη σύνδεση Βερολίνου Μπρεσλάου και ενώ στο πολωνικό κομμάτι έχει ήδη κατασκευαστεί το, το έργο, στη γερμανική πλευρά δεν έχει χτιστεί, δεν έχει κατασκευαστεί αυτή η γραμμή. Μπορείτε να εγγυηθείτε εσείς ότι θα χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο, γιατί θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, γιατί θα υπηρετήσει το, το, το στόχους για το κλίμα. Και ακούμε ένα όχι. Και εδώ κάνατε ένα, φοβε... ένα εξαιρετικό κατάλογο. 127 δισεκατομμύρια αξίζουν τα έργα, τα 63 από αυτά ε, αφορούν αυτοκινητοδρόμους. Δεν έχω ακούσει ούτε έναν επιστήμονο να δηλώνει ότι με νέους αυτοκινητοδρόμους θα υπηρετηθούν οι στόχοι για το ε, κλίμα. Υπόθηκε και από έναν επιστήμονα τη δεκαετία του 70 ότι όποιος σπέρνει δρόμους θερίζει κυκλοφορία στους δρόμους. Και σε κάθε περίπτωση, αν η, ευρωπαϊκή, η γερμανική κυβέρνηση ετηθεί ένα νέο έργο, θα πρέπει εσείς να πείτε όχι. Γιατί ο Υπουργό ε, Συγκοινωνιών είπε ότι χρειάζονται 7 δισεκατομμύρια ετησίως για τη συντήρηση των υποδομών στη Γερμανία. Είμαι την προηγούμενη εβδομάδα σε σύνοδο στο Παρίσι υποστηρικτών των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι είπαν ότι ο βασικότερος στόχος μας θα πρέπει να είναι η συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Κανονικά δηλαδή θα πρέπει να, πούμε, να πείτε στη Γερμανία δεν θα γίνουν νέα έργα. Δείτε πώς και αν μπορείτε να συντηρήσετε τις υπάρχουσες υποδομές. Υπάρχουν υποδομές που δεν χρησιμοποιούνται πια στη Γερμανία γιατί δεν έχουν συντηρηθεί. Και τέλος. Αναφέρθηκε αυτοκινητόδρομος Ρον ε, Τωρίνο. 80 χιλιόμετρα νέες σύραγγες. Άντε ξανά να τρυπήσουμε τις, τις Άλπεις. Πόσες θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν. Πόσο θα, θα υπάρξει, πόσο θα συμβάλλει αυτό το έργο στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα. Ποιες δυνατότητες βλέπετε να μπορούμε να πούμε όχι αυτό το έργο αντιτίθεται και στους τρεις στόχους του σχεδίου ε, Juncker θα προτείνουμε κάτι εναλλακτικό. Αν θέλετε εναλλακτικέ λύσει, ελάτε σε εμά. 100-200 έργα θα σα προτείνουμε. Αλλά όχι 500 δισεκατομμύρια, γιατί τέτοιου είδου έργα μπορεί να γινει μονο μόνο 2-3. Και πώ, το ερώτημα είναι, πώ μπορείτε εσεί να κατευθύνετε με βάση μια τέτοια λογική τα όσα θα συμβούν στο μέλλον. Αυτή είναι η συζήτηση που έχουμε κάνει πολλέ φορέ. Την κάναμε και χτε, την κάναμε και σήμερα και νομίζω ότι θα την ε, κάνουμε και στο μέλλον αρκετέ φορέ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κριστόφερσον. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι εμείς οι τρεις δεν μπορούμε προφανώς να επιβάλλουμε τίποτα. Δεν αποτελεί τμήμα της εντολής μας. Δεν μπορούμε εμείς να διαμεσολαβήσουμε. Δεν μπορούμε εμείς να, μπορούμε να, να προσδιορίσουμε προβλήματα που πρέπει να επιληθούν αν θέλουμε ε, να υλοποιηθούν ορισμένα έργα με, το... με τον κατάλληλο τρόπο. Αλλά για η απόφαση για την επίλυση των προβλημάτων αυτών θα πρέπει να ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Δεν είμαι όμως τόσο απεσιόδοξος. Αν δείτε τη στρατηγική για την ενιαία αγορά, θα δείτε ότι έχουν αρθεί χιλιάδες εμπόδια. Έχουμε ένα πολύ πιο ε, φιλελεύθερο, απελευθερωμένο ε, οικονομικό σύστημα σήμερα από ότι το 1985. Άρα μπορεί να γίνει. Ορισμένα ε, εμπόδια όμως έχουν εθνικό χαρακτήρα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει και να επιλύσει προβλήματα. Αλλά αυτό αφορά αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών. Σε, όσο, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να αναλάβουμε δράσεις στις κρατικές χορηγήσεις, στις, ε, στα, στις προδιαγραμμές, στα πρότυπα. Έχουμε Άρη σε επίπεδο ένωσης πολλά εμπόδια. Υπάρχουν όμως κάποια εθνικά εμπόδια όπου τα κράτη-μέλη επιμένουν ότι η Ένωση δεν θα πρέπει να έχει καμία συμμετοχή. Κρίμα είναι, αλλά έτσι είναι. Και συμφωνώ με τον Πρόεδρο απολύτως ότι υπάρχουν πολλά κενά στο σύστημα υποδομών. Όταν πηγαίνω από την Αλσατία στην Γερμανία, λείπουν ακόμη 15 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου που να συνδέουν τον γερμανικό με τον γαλλικό ε, με τον, γαλλικό, τον γερμανικό με τον γαλλικό αυτοκινητόδρομο. Υπάρχει μόνο ένας αυτοκινητόδρομος που συνδέει τους, τους, τα δύο συστήματα αυτοκινητοδρόμων της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ε, καμία σχέση βεβαίως όταν ε, συγκρίνω τη σύνδεση με αυτοκινητόδρομο μεταξύ Βελγίου και Ολλανδίας ή Βελγίου και Γερμανίας. Σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα είναι ότι πολλά εμπόδια έχουν ήδη αρθεί και μπορούν να αρθούν και σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε. για ποιο λόγο πρέπει να ενδιαφέρονται τα συντεξιδοτικά ταμεία και τέτοιου είδους οργανισμοί στις ε, επενδύσεις υποδομών. Εγώ γνωρίζω τέτοια ταμεία που ε, που ε, χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά στο γαλλικό σύστημα αυτοκινητοδρόμων γιατί οι ιδιοκτήτες έχουν αγοράσει λιμάνια, έχουν αγοράσει ε, αεροδρόμια ε, στη Δανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε άλλες ε, χώρες. Στο παρελθόν τα συνταξιδοτικά ταμεία επένδυαν για παράδειγμα στη δασοκομεία δεν το κάνουν πια τόσο πολύ, αλλά πάντοτε ψάχνουν επενδυτικές ευκαιρίες με καλή απόδοση. Το προφίλ για την εξοικονόμηση στα συνταξιδοτικά ταμεία είναι πολύ συχνά το ίδιο με το προφίλ της εξοικονόμησης σε επενδύσεις για τις υποδομές. 4-5 χρόνια για παράδειγμα η πρώτη απόδοση επένδυσης. μία 4% αύξηση ε, στο παρελθόν είχε σαν αποτέλεσμα ε, αύξηση ε, των, κερδών για όσους συμμετείχαν σε αυτά τα συνταξιδοτικά ταμεία. Αλλά φέτος τι γίνεται στη Γερμανία για παράδειγμα. Γιατί πολλά συνταξιδοτικά ταμεία πλέον είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποσχέσεις και στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Υπάρχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το εποπτικό συμβούλιο μιας ε, εταιρείας συνταξιοδοτική ε, δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση αποτυχίας μιας επένδυσης. Ε, έχουν όμως μία νομική ευθύνη να τηρήσουν τις ε, δεσμεύσεις τους, διαφορετικά μπορεί να βρεθούν στη φυλακή. Και δεν είναι παρκές να μας λένε «Α, ε, μαζί της ε, το το Υπουργείο Οικονομικών ε, να κάνουν. Ε, έχουμε έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για αυτό το θέμα, η οποία είναι πολύ πιο δραστήρια σήμερα στην αξιολόγηση της ποιότητας των προγραμμάτων ε, από ό,τι 5-10 χρόνια πριν. Αυτό βέβαια σημαίνει πρόοδο αλλά είμαι βέβαιος ότι οι ασφαλιστικές και οι εταιρείες και οι συνταξιοδοτικές εταιρείες ε, ε, εξακολουθούν να αναζητούν πολύ μεγάλη απόδοση. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από την αποδοτικότητα του προγράμματος 5, 6, 7% άμα είναι πάρα πολύ ψηλή και κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο κακό αυτό γιατί συχνά η εναλλακτική είναι να μην εφαρμοστεί ποτέ το πρόγραμμα. Αυτή είναι η εναλλακτική επιλογή σε πολλά πολλά κράτη-μέλη. Αν δεν υπάρχουν ιδιωτικοί επενδυτές, ιδιώτες επενδυτές, δεν θα, εξαφανιστούν τα προγράμματα. Είναι ελεύθερη επιλογή, αλλά πρέπει να το ξέρουμε ότι μπορεί αυτές να είναι οι συνέπειες. Με ρωτήσατε επίσης πόσα χρήματα υπάρχουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ε, είχαμε πει... Ε, υπάρχουν προγράμματα που θα τύχουν ιδιωτική επένδυση και προγράμματα στα οποία οι ιδιώτε επενδυτέ θα πούνε δεν μα ενδιαφέρουν, δεν μας ενδιαφέρει να επενδύσουμε σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό στη Στουτγάρδη ε, ή κάπου στο Βερολίνο. Α, το ξέρετε, αυτό λέει ο πρόεδρο. Ναι, διαβάζω τις γερμανικές εφημερίδες, λέει ο κύριο Χριστόφερσεν. Τέλος πάντων, λίγα ακόμα πράγματα θα ήθελα να πω. Η συγκέντρωση των προγραμμάτων. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Φιλανδία, Εσθονία ε, σχεδιάζουν ε, να οικοδομήσουν ένα σταθμό ε, υγροποιημένου αερίου και να το συνδέσουν με έναν αγωγό που θα πηγαίνει σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ναι, ένα συνδυασμός, ας το πούμε έτσι, προγραμμάτων. Υπάρχει και κοινή επιδότηση. Αν, αν αν ας πούμε αν θέλουμε να συνδέσουμε δύο ε, πόλεις ε, πρέπει πρέπει να ε, προβλεφθεί για ένας αυτοκινητόδρομος και ένα τμήμα των εσόδων των αυτοκινητοδρόμων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ε, χρηματοδοτηθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά το θέμα είναι πόσο πιο μακριά μπορεί να πάει κανείς με, αυτή την, με αυτό το συνδυασμό χρηματοδότης και το συνδυασμό των επιδοτήσεων για τους ξένους επενδυτές. Ναι, βεβαίως θα μιλήσουμε με τους Νορβηγούς και το, ε, το, το Norwegian Petroleum Fund. Ναι, βεβαίως θα μιλήσουμε, θα δείξουμε καμιά ματιά στην αγορά να δούμε κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον και βέβαια οι υπεύθυνοι λήψη αποφάσεων θα αποφασίσουν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Μπορεί να βρούμε για παράδειγμα ότι υπάρχει μια ευκαιρία στο ένα ή στο άλλο, μία στην άλλη επένδυση και να ολοκληρώσω λέγοντας ένα μόνο πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να απαντήσουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Είμαστε ακόμη σε μία φάση που ακούμε και προσπαθούμε να ε, συγκεντρώσουμε γνώσεις και εμπειρίες Ακούμε αυτά που μας λέτε κι εσείς και αυτό θα έχει ένα σημαντικό αντίκτυπο στο πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά μας. Εμένα το σουηδικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι είμαι μισό σουηδός, δεν με εντυπωσιάζει να σας πω την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικό, αλλά αυτό τέλος πάντων είναι άλλο θέμα. Ευχαριστώ, Κουρτ Μπόντεβιλ. Έως το 2030 χρειάζονται 600 δισεκατομμύρια, τα επόμενα 7, 26. Άρα χρειαζόμαστε άλλες λύσεις. Υπάρχουν κανονισμοί για το TNT και για το CEF που θέτουν συγκεκριμένες ε, με συγκεκριμένα κριτήρια. συνοριακά έργα, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αυτά τα 26 δισεκατομμύρια θα πρέπει να προσανατολιστούν με βάση αυτά τα κριτήρια που δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω άλλων πηγών. Αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικότερα ε, έργα, καθήκοντα της ε, Γενικής Διεύθυνσης MOVE σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Αλλά για τα υπόλοιπα κεφάλαια που μπορούν να κινητοποιηθούν υπάρχουν όντως κάποιες, ε, κάποια εμπόδια. Θα πρέπει δηλαδή ε, στη Eurostat να συμπεριλάβουμε ότι δεν υπάρχουν μόνο τα κόστη κατασκευής αλλά και συντήρησης και λειτουργίας. Χρειαζόμαστε κανόνες που θα είναι πιο απλοί, που θα διευκολύνουν το έργο μας και για τα κριτήρια Μάστριχτ στο EFSI είναι αυτονόητο ότι τα χρήματα, τα κονδύλια ε, του EFSI δεν θα, ε, ε, δεν θα ανταποκρίνονται στα κριτήρια του Μάστριχτ υπάρχει διάκριση μεταξύ έργων που, θα, που είναι απαραίτητα για την κοινωνία που, και έργων που είναι κερδοφόρα στο πρώτο έγγραφο είχαμε καταστήσει σαφές ότι η χρηματοδότηση από τους χρήστες είναι ένα από τα εργαλεία που πρέπει να συνδυαστεί με άλλα. Αλλά αυτό το εργαλείο θα υπάρχει στους δρόμους κατά κύριο λόγο. Θα υπάρχουν διόδια θα, ε, τα οποία θα αποφέρουν κέρδη για, πιθανώς, ε, για πιθανούς επενδυτές. Κάτι τέτοιο όμως αποκλείεται στην, ε, στις πλωτές οδούς και στους σιδηροδρόμους. Και στα αεροδρόμια ενδεχομένως να μπορεί να ε, εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, αλλά στους σιδηροδρόμους θα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Γι' αυτό το λόγο το 80% των ε, κονδυλίων ε, του CEF κατευθύνονται στις, ε, στις, στους σιδηροδρόμους. Και να πω και για το ερώτημα, επειδή τέθηκε το ερώτημα. Κατά έργο βεβαίως θα υπάρχουν συγκεκριμένα χρωματοδοτικά συστήματα. Θα πρέπει να εξετάζουμε ποιες είναι οι ε, απαιτήσει τη ισχύ στην κάθε χώρα. Και τέλος, οικολογικό αποτύπωμα. Ναι, αλλά αυτό υπάρχει ίδιο κριτήριο σε κάθε έργο του CEF, αφού ήταν άλλωστε και τμήμα ε, του έργου ελέγχου μας, του ελεγκτικού μας έργου. Άρα από τη στιγμή που ένα έργο μπαίνει μέσα σε αυτό το pipeline, σε αυτόν τον αγωγό έργων, θα πρέπει να πληρεί και ορισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια. Άρα αυτό το κριτήριο περιλαμβάνεται ήδη. Και τέλος, όλες οι προβλέψεις για τις ε, μεταφορές έχουν, ε, έχουν ήδη ε, υπερβαθεί. Αυτό που ε, πρόκειται να συμβεί στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ε, θα είναι καταστροφικό. Γι' αυτό δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην πραγματικότητα μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Αντίθετα, υπάρχει ανάγκη ε, συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Για τις θέσεις απασχόλησης υπάρχουν δύο επίπεδα. Αφενός υπάρχουν οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούν το που δημιουργεί το κάθε έργα έργο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και θέσει απασχόληση που ε, δημιουργούνται έμεσα στην ε, κάθε τοποθεσία. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι για τρία χρόνια όσο θα χτίζεται το τάδε έργο να δημιουργηθούν αυτές και αυτές οι θέσεις ε, απασχόλησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σέκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από ό,τι κατάλαβα ξεπεράσαμε το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας και πολλά σημεία που θέσατε ε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Εκαλύφθησαν πολλά σημεία από τους συναδέλφους. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν θα είμαι λακωνικός. Θα αναφερθώ σε δύο ή τρία γενικά θέματα. Πρώτα απ' όλα αυτό που έθεσε ο κ. Βάντερ Κάμπ για τη συμπράξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είπε ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ότι αυτές οι συμπράξεις αποδίδουν κάποια αξία. Έχω αντίθετη άποψη. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις προσφάτως αλλά και παλαιότερα. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια σχετικά στοιχεία στην τελική έκθεση, αν συμφωνούν οι συνάδελφοι. Πιο συγκεκριμένα για την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η οποία μπορεί να αποδειχθεί άκρος επωφελής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, τον εφοδιασμό, την τήρηση χρονοδιαγράμματων, την ποιότητα ε, του έργου, ε, μια προσέγγιση κύκλου ζωής κλπ. Αυτό θα το τονίσουμε γενικότερα η χρηματοδότηση των υποδομών είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουν οι φοιτητέ μου γιατί είναι ένα παράδειγμα αποτυχίας της αγοράς. Τα μηνύματα των αγορών για τη διανομή, για την κατανομή των πόρων, κυρίως των χρηματοπιστωτικών, οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα, δηλαδή αυτοκινητόδρομοι, εντύσεις σιδηροδρόμων κλπ η καλή πολιτική απόφαση πρέπει να προσπαθεί να παρεμβαίνει άμεσα όπως το CEF ή κυβερνητικής χρηματοδοτήσεως υποδομών είτε να γίνεται διόρθωση των αποτυχιών της αγοράς. Ένα παράδειγμα ήδη αναφέρθηκε. Θετική αρνητική συνεισφορά όσον αφορά το περιβάλλον. Αυτό δεν λαμβάνεται κανονικά υπόψη στην περίπτωση των σιδηροδρόμων, διότι εκαλύπτονται οικονομικά από το κράτος και δεν γινόταν ο δέον υπολογισμός. Αν πρέπει να γίνει προσφυγή στην αγορά πρέπει να υπάρχει σωστή προσέγγιση και να ληφθεί υπόψη η νέα κατάσταση και όχι παλιά, γιατί η κατάσταση τώρα είναι καινούργια. Είναι θέμα κινήτρων. Το είπε και ο κύριος Τζιλ, από ό,τι κατάλαβα το θέμα αυτό. Έχουμε το μοντέλο το ε, ελβετικό. Υπάρχουν σαφή κίνητρα και αντικίνητρα που κινούν τις επενδύσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με την πολιτική απόφαση. Και διασταυρούμενη χρηματοδότηση βρίσκει απάντηση εδώ. Η διασταυρούμενη χρηματοδότηση, εάν εφαρμοστεί σωστά, είναι ένας τρόπος να εξετάζει κανείς διάφορα έργα σαν πακέτα. Αν υπάρχουν Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά εμπόδια, μέσω διασταυρούμενης χρηματοδοτήσεως βρίσκεται μια λύση που παράγει καλύτερη ισορροπία παρά να αφήνει τα πάντα να ρυθμίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς. Κανονισμός, φερεγγιότητα 2 κλπ. Το άλλο θέμα που εφήγει. Σημαντικότατοι κανόνες. Θεσπίστηκαν ούτω ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του κινδύνου. και να διοχετεύονται πόροι για τη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα. Κάτι που δεν γίνεται ανοιχτά αποδεκτό, έχοντα υπόψη ότι μετά δημόσιο τομέα θα χρηματοδοτεί υποδομέ και ούτω καθεξής. Αυτό είναι τυπικό του Solvency 2. Εάν θέλει κανείς πολύ χαμηλό κίνδυνο δεν πάει πουθενά. Πρέπει να αποδεχθεί κανείς υψηλότερο κίνδυνο. Αν συνεχιστεί η διοχέτευση πόρων προς το κράτος και το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις, πάλι δεν πας πουθενά. Γι' αυτό, επειδή το πλαίσιο είναι εντελώς διαφορετικό, σε σύγκριση του όταν αποφασίστηκαν και σχεδιάστηκαν το Φερεγγιώτητα 2 και η Βασιλεία 3 πρέπει να επανεξετάσουμε τα πράγματα από το 0 και να βρούμε ένα νέο πλαίσιο που είναι προσαρμοσμένο στις σημερινές ε, εποχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό της σημερινή διάταξη. Ευχαριστώ και τους τρεις κυρίους για τις παρουσιάσεις τους. Και με αυτό... Περνάμε στα διάφορα, στο επόμενο θέμα δηλαδή τη ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι 16 Μαρτίου στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ και γεια σας.